Euh, Σημείο 1 της ημερησίας διάταξης. Έγκριση της ημερησίας διάταξης. Σας έχει διανεμηθεί το σχέδιο ημερησίας διάταξης το οποίο και εγκρίνεται. Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ο συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Επομένως να χαμογελάτε να παίρνετε το λόγο. Δεύτερη ανακοίνωση. Στο φάκελό σας θα βρείτε την ανακοίνωση που προτίμασε η Γραμματεία όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την συζήτηση που θα έχουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το οποίο θα συζητήσουμε στην, στο δεύτερο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης, σημείο 3 τροποποίηση του κανονισμού για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής. Πρόκειται για ένα σημαντικό κείμενο. Θα εξετάσουμε γι' αυτό λοιπόν τις τροπολογίες, 24 στο αριθμό, οι οποίες υπευλήθησαν για την έκθεση λοιπόν αυτή από τον κύριο Καρμπνόχα, μάλλον για την έκθεση του κύριου Καρπνό, ο οποιο ε, υπέβαλε αρχικά 17. Κύριε εισηγητά, έχετε τον λόγο. Δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι και όλοι εισηγητές για την έκθεση αυτή. Ελπίζω οι εργαζόμενοι στις πολιτικές ομάδες να τους ειδοποιήσουν προκειμένου να έρθουν εδώ πέρα και να λάβουν το λόγο. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από την ψηφοφορία αύριο πρέπει να δούμε 24 ε, τροπολογίες και από ό,τι μαθαίνω 4 ή 5 έχουν αποσυρθεί από τις αρχικές. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου θα καταψηφίσουμε, θα προτείνω δύο καταψηφίσεις του, του Αντιπροέδρου Τόμας Μαν. Όλες οι άλλες τροπολογίες, ε, όλες τις άλλες τροπολογίες θα τις υποστηρίξω. Ως προς τις ε, τροπολογίες του κυρίου Μαν, αυτές είναι καθαρά συντακτικές. Γι' αυτό θα ήθελα να τις αποσύρει η δυνατόν και στη συνέχεια με καθαρή τη συνείδηση θα μπορέσω να υποστηρίξω τις υπόλοιπες και σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Ε, Κυρία Ισάια, ευχαριστώ. Ο εισηγητής ακολουθεί τη θέση του Συμβουλίου εκ του Σύνεγγης, γι' αυτό δεν έχω να αντιτάξω κάτι μόνο για την 27. Η τροπολογία 27 δεν ξέρω κατά πόσο έχει αποσυρθεί ή όχι. Εκεί έχουμε ένα θέμα ίσον σημασία. Α, εντάξει, έχει αποσυρθεί. Εντάξει, εντάξει, από τη δική μας πλευρά τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Οβίρ, η κυρία Οβίρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τους ε, φιλελευθέρους. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την ε, εντάχει, την εργασία που διεκπαιρεώθηκε μάλλον τάχιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γιατί όπως ξέρουμε όταν πρόκειται για κανονισμό δεν μπορεί παρά να αντικατασταθεί από άλλο κανονισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συμφωνήσουμε. Όπως είπε και ο Μίλαν, υπάρχουν τροπολογίες που ε, μερικές δεν θα τις υποστηρίξουμε και οι άλλες συμβαδίζουν με αυτά που συζητήσαμε στο Συμβούλιο. Ως προσυντακτικά θέματα δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε δηλαδή οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές. Θα υποστηρίξουμε τον κανονισμό αύριο κατά την ψηφοφορία. Ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μίλαν, έχουμε συνήθως ίδιες ιδέες και λες ε, πως ε, θα μπορούσα να αποσύρω το μου. Όσον αφορά την υπαριθμόν 29, νομίζω πως ε, το ζήτημα είναι απλά γλωσσικό. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, νομίζω πως είναι ταυτόσιμο με το προηγούμενο. Και μετά αντί δεις την υπαριθμόν 17 και τη συγκρίνεις με την 18 της κυρίας Γιούτα Στάινρουπ, νομίζω πως είναι ταυτόσιμες. Αν λες πως συμφωνείς με τη 18 της Γιούτα και εμένα δεν απέχει πολύ να την αποσύρω τη 17 υπέρ της τροπολογίας της ε, κυρίας Γιούτα Στάινγκοφ. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου επί της 18, την οποία εγώ βρίσκω μια χαρά ούτως ή άλλως. Οπότε, Μίλαν, μπορείς να μας να το ξεκαθαρίσεις γιατί και στο 2 ε, νομίζω συμφωνούμε αν και τα τον τον εργαζομένων θα τα δούμε. Ε, Ευχαριστώ. Ήδη συζητήσαμε αυτό το θέμα αρκετές φορές. Όπως ξέρει ο εισηγητής, εμείς οι σοσιαλιστές είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία του, διότι καλύπτει τις βασικές μας ανησυχίες και έχουν υποβληθεί και τροπολογίες. Και από όσο βλέπω καταπίπτουν καταρχήν οι 18 και οι άλλες συναφείς και έτσι νομίζω ότι επιλύονται δύο βασικά ζητήματα. Ε, καταρχήν ως προς τους εργαζομένους της αεροναυσιπλοείας που τώρα πλέον δεν πλήττονται με βάση τις ε, δραστηριότητες όπως τις προτείνουμε γιατί υπάρχει και νομική ασφάλεια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτουμε το θέμα της ε, κοινωνικής ασφάλισης. Και επιλύονται και τα θέματα των ε, διασυνοριακών εργαζομένων. Γι' αυτό θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες του κυρίου Κάμπρνοχ, έτσι ώστε αυτή η νομοθεσία να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση. Euh, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Επιτροπή σας για την πολύ γρήγορη εργασία που κάνατε και ελπίζουμε κι εμείς ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Με Αυτό είναι πολύ σημαντικό, για τους πολίτες αυτούς οι οποίοι καλύπτονται από την τροποποίηση του κανονισμού που έχουμε εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη, θα πάρετε πάλι το λόγο. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για το ότι μου δίνετε δύο φορές το λόγο. Μόλις μίλησα με την κυρία Στάινρουκ. Απέσυρε την υπαριθμόν 18 Οπότε δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Αλλά την κοίταξα, κοίταξα τη 16. Η δικιά μου 17 είναι η ίδια με την 16. Οπότε καταπίπτει αυτομάτως γιατί είναι πολύ παρόμοιο με αυτό το οποίο έχει κάνει. Γι' αυτό ήθελα το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Μετά, στο σημείο 29. Το 28 δεν απέχει πάρα πολύ από το 29 είναι οριακά γλωσσικά ζητήματα. Οπότε αν γράφει καταπίπτει ή αν υιοθετηθεί δεν είναι πρόβλημα. Οπότε αν ε, υιοθετηθούν όπως είναι αυτές οι τροπολογίες, τους ή άλλως η τοποθέτηση ε, έχει υιοθετηθεί. Αυτά και ευχαριστώ. Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, δεν αποσύρεται τις τροπολογίες, αλλά θα καταπέσουν αν περάσουν αυτές του εισηγητή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι τροπολογίες σας δεν θα απέχουν πολύ από το κείμενο του εισηγητή. Θα δούμε λοιπόν ε, και την αρρύθμιση που θα γίνει στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ποια είναι η σειρά που θα ακολουθήσουμε. Θα δώσουμε πάλι το λόγο στον εισηγητή Πάντως στην συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφύγουμε, να επαναλάβουμε κάποιες συζητήσεις που ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα. Όταν η συγητής αναφερθεί μάλλον ότι είναι συγητή αναφέρεται πολύ συχνά στα όσα έχουν συμφωνηθεί με του κοιόδη συγητέ. Πολλοί από εμά δεν γνωρίζουμε ακριβώ τι έχει συμφωνηθεί. Μα απασχολεί ιδιαίτερα λοιπόν η νομοθεσία αυτή και θα έπρεπε κάποια στιγμή κάποιο να εξηγήσει σε όλου του συναδέλφου τι διακυβεύεται με την προτινόμενη αυτή νομοθεσία, τι αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων όχι και κλεισμένων των θυρών αναγκαστικά, αλλά συζητήσεις οι οποίες δεν γίνανε, αν θέλετε, στην ολομέλη εδώ της Επιτροπής μας. Θα ήταν σημαντικό να μας πείτε κάποια στιγμή ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία της διαπραγμάτευσης, ποια ήταν τα σημεία εκείνα στα οποία το Συμβούλιο επιθυμούσε να γίνουν κάποιες προσαρμογές και να μας εξηγήσετε επίσης και ποια είναι η τοποθέτηση όλων των συμβαλωμένων μέρων στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση. Συγγνώμη που απευθύνομαι σε εσά κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι σε ένα γενικότερο πνεύμα διαφάνεια είναι καλύτερα να μα εξηγήσετε τα πράγματα που να μα λέτε απλώ ότι συμφωνήσαμε με του κοιόδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι μπορώ να πω πως δεν άλλαξε τίποτα σημαντικό στην πρόταση από την πρώτη φορά που τη συζητήσαμε, οπότε μπορώ να επαναλάβω αυτά τα οποία είχα πει τότε. Οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, έχουμε τα κριτήρια στην περίπτωση που συγκεκριμένο άτομο δεν εκπληρώνει ουσιαστικό τμήμα των δραστηριοτήτων του σε ένα μόνο κράτο μέλο, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη. Έτσι είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί κάποιο να ζει σε μια χώρα και να εργάζεται σε άλλη ή να εργάζεται σε πολλέ χώρες και να μένει σε μία από αυτές. Η πρότασή μας προβλέπει σαφείς ορισμούς για το τι κάνουμε σε διάφορετικές περιπτώσεις. Ειδικά αυτό ισχύει και για τους ε, διασυνοριακά εργαζόμενους. Ένας άλλος τομέας είναι ο καθορισμός του τόπου της έδρας των εταιριών. Ε, ειδικά όταν μιλάμε για πληρώματα αεροπλάνων. Ήταν δύσκολο να πούμε πού υφίσταται η έδρα των ε, πληρωμάτων αεροπλάνων οπότε συμφωνήσαμε σε αυτό το οποίο συμφώνησε και το Συμβούλιο δηλαδή το κριτήριο κατοικίας και το κριτήριο μου συγχωρείτε της ε, βάσης ε, εκεί όπου προσγειώνονται περισσότερο ή από εκεί από όπου απογειώνονται συχνότερα ή εκεί όπου κατοικούν. Και ο τρίτος τομέας επιδόματα ανεργίας για δύο συνεργατικούς εργαζόμενους. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους. Ε, διαφορετικά κράτη-μέλη βεβαίως έχουν διαφορετική νομοθεσία που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μετά τελειώνουν τη δουλειά τους και επιστρέφουν στο κράτος μέλος κατοικίας. Και το ερώτημα είναι από πού παίρνουν επίδομα ανεργίας, εάν παίρνουν. Σε κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρο, Λετωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανεργία των ελευθέρων επαγγελματιών. Σε άλλες χώρες υπάρχει. Οπότε το είδαμε αυτό το ζήτημα, προτείναμε μια λύση για δύο χρόνια και μετά θα το αναθεωρήσουμε. Συναντήσαμε επίσης εκπροσώπους της Προεδρίας πολλές φορές τους σκιώδεις εισηγητές και ξεκαθαρίσαμε διάφορα πράγματα. Η νομοθεσία αυτή είναι τεχνική, γι' αυτό χαίρομαι για το ότι με τη βοήθεια της Γραμματείας Επιτροπής μπορέσαμε να προετοιμάσουμε μια πρόταση την οποία ελπίζω να στηρίξουν όλοι. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τις συναντήσεις μας με την Δανική Προεδρία είδαμε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και η κοινωνική νομοθεσία που θα αποφασιστεί. Γι' αυτό οι συζητήσεις που έγιναν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι αρκετά θετικό. Γιατί υπάρχει ευρεία συνένεση από ό,τι φαίνεται. Άρα αύριο θα ψηφίσουμε έτσι ώστε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο να αποφασίσουμε και εμείς και η Προεδρία της Δανίας, αν όλα πάνε κατευχήν. Προχωράμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στην κυρία Ζούμπερ για να εξετάσουμε την έκθεσή της για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών που θα είναι το 2013 και όχι το 2014 που έχουμε εμείς εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ως προς τη γνωμοδότησή μας λάβαμε πολλές τροπολογίες, πάνω από 90, και με βάση μία συζήτηση που έγινε, μία διευρυμένη συζήτηση, φτάσαμε σε 11 προτάσεις συμβιβασμού, αν δεν κάνω λάθος. Κατά τη γνώμη μου, στην ουσία αναβαθμίζουμε τον κανονισμό γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις, να τις καταπολεμήσουμε ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιώματα ηθαγένειας που συμπεριλαμβάνουν και κοινωνικής φύσης ε, δικαιώματα που θα πρέπει να εγγυηθούμε σε κατοίκους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις προτάσεις συμβασμού, έχει ως εξής θα πρέπει το Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με την ελεύθερη κυκλοφορία να ασχοληθεί και με το θέμα καταπολέμησης των διακρίσεων έτσι ώστε να μην έχουμε φτηνή εργατική δύναμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης καθώς και στα μέλη της Γραμματείας. Ευχαριστώ πολύ. Steinrück. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εκπροσωπώ την κυρία Μπίρκετ Σίπελ, η οποία κολλείεται και θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγκήτρια για το ότι καταφέραμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις, τις οποίες υποστηρίζουμε όλες εμείς οι σοσιαλδημοκράτες. Βρήκαμε ε, συμβασμούς για ζητήματα μη ε, διάκρισης, ενημέρωσης όλων των πολιτών, καθώς επίσης και τη σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς για ενίσχυση των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών ήταν κάτι το οποίο πέρασε. Κρίμα θεωρεί η κυρία Σίπελ πως για κάποια θέματα οι συμβασμοί δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο θα ήθελε ε, ειδικά για κάποιες ευπαθείς ομάδες ε, για να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε και να τις ενημερώσουμε τα προβλήματα των Ρωμά, αποσπασμένων, εργαζομένων τα οποία δυστυχώς δεν αναφέρονται τόσο ρητός ε, πλέον. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες μπορούμε να στηρίξουμε αυτό τον συμβασμό. Και εξ ονόματος συναδέλφου, σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Ja, ich möchte auch herzlichen Dank sagen, Frau Zuber, für die äh, äh Leitung äh, dieses Prozesses. Der Κύριος Becker. Σα ευχαριστώ. Νομίζω πως ήταν ένα πάρα πολύ καλός συμβιβασμό και δίκαιος για το θέμα. Αγγίζει και το θέμα της ευρωπαϊκής υπηκότητα και της συμμετοχής των ιδίων των πολιτών. Ένα περίπλοκο θέμα. Και βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ε, ε και απόψει που λύθηκαν με τρόπο επαγγελματικό και φιλικό. και θα ήθελα άρα να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε εδώ πέρα και η επικοινωνία αυτού του θέματος στους πολίτες είναι το σημαντικότερο. Γιατί ο πολίτης πρέπει να ενημερωθεί για αυτά τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχει. Και αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε και πρέπει να τα αναλάβουμε. Ευχαριστώ. Ε, Μαρκίν και κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε Καταφέραμε τελικά με τον έναν άλλο τρόπο να καταλήξουμε στις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Έχουμε κάποιες πάρα πολύ καλές ιδέες. Πρόκειται για μια έκθεση ιδιαίτερα προδραστική. Θα μας επιτρέψει πραγματικά να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι τα δικαιώματά τους και νομίζω ότι μας δίνεται και μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως είπε και ο προλαλής σας, για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να καταλάβουν καλύτερα τα ωφέλη του να είναι κανείς πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εισαγήτρια. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε κάποιες καλές α, λογικές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Παδοπούλου έχει τώρα το λόγο και η Μάκιντήρη συνέχεια. Ευχαριστώ. ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια εγώ είμαι συγγήτρια για την Επιτροπή Ελευθεριών και μάλιστα οι περισσότερες τροπολογίες ε, συμφωνούν με τις προτάσεις μου. Αλλά θα ήθελα να θέσω κάτι, γιατί όπως ξέρετε του χρόνου θα έχουμε την 20η επέτειο της ε, αναφοράς στη συνθήκη του Μάστριχτ στην ευρωπαϊκή υπηκότητα. Και όταν το 2010 είχαμε την ε, αναφορά για την έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιήθηκε ο τίτλος υπηκότητα αντί για πολίτες. Οπότε αντί για ευρωπαϊκό έτος των πολιτών θεωρώ πως θα έπρεπε να λέμε ευρωπαϊκό έτος υπηκότητας. Είναι σημαντικό αυτό γιατί συζητάμε για την ανάγκη να αυξηθεί η ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών, να ξέρουν τι είναι αυτή η ευρωπαϊκή υπηκότητα και θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα δικαιώματα, ελεύθερη διακίνηση, ε, εργασία χωρίς διακρίσεις, αλλά και άλλα δικαιώματα που προέκυψαν, προκύπτουν από αυτή την επικότητα. Και σας παρακαλώ να σκεφτείτε την ιδέα να αλλάξετε τον τίτλο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι πως ο προϋπολογισμός για φέτος είναι μόλις ένα εκατομμύριο σε σύγκριση με τα 27 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια που έχουν άλλα ευρωπαϊκά έτη. Οπότε είναι cannot... παρόλες καλές προθέσεις και εκθέσεις, αν δεν υπάρχουν λεφτά δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες για τα δικαιώματα και τα εμπόδια και τις υποχρεώσεις που έχουν. Αυτά και παρακαλώ να σκεφτείτε αυτό που είπα. Κυρία Μακιντάιρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναγνωρίζω πως κάποιοι θεωρούν πως το 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά λεφτά αλλά εγώ αμφισβητώ το κατά πόσον είναι κατάλληλη αυτή η πρόταση. Ε, αν δει κανείς τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, τον κόσμο που υποφέρει από τη λιτότητα, στην Πορτογαλία με το ε, επίπεδο ανεργίας, ε, ο κόσμος θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα είναι άσχετα, δεν αναγνωρίζουν το τι σημαίνει να είναι κανείς σήμερα πολίτης στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ πώ δεν πρέπει να ξοδεύουμε λεφτά λοιπόν καθόλου για τέτοια πράγματα. Ε, ειδικά αυτή τη στιγμή. Ε, αφού τα ξοδεύουμε όμως, νομίζω πως χάνουμε και κάποιες ευκαιρίες. Κάτι το οποίο με λυπεί και θα με έχετε ξανακούσει οπωσδήποτε να το λέω, είναι πως μιλάμε για δικαιώματα, αλλά δεν μιλάμε για υποχρεώσεις. Ξέρετε αυτά είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Οπότε για να είναι κάποιος πολίτης πρέπει να αντιλαμβάνεται και τις ευθύνες του και όχι μόνο τα δικαιώματά του. Και αυτό δεν αναφέρεται καθόλου στην έκθεση και στην ε, Επιτροπή Ελευθεριών το ίδιο. Επίσης θεωρώ πως χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη γιατί περισσότεροι θεωρούν πως είναι πολίτες μιας χώρας συγκεκριμένης. Πολύ πριν, εάν κιόλα θεωρήσουν ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το σημαντικό είναι να ενθαρρύνουμε την υπηκότητα. Εάν εγώ είμαι όπως αισθάνομαι Βρετανίδα ή ο καθένας οποιασδήποτε χώρας, η υπηκότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενθαρρύνεται και πρέπει να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, την ανάληψη ευθυνών και θεωρώ πως ολόκληρη αυτή η έκθεση της Κομισιόν και η απάντηση και η αντίδραση νομίζω ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Ο κύριος Μαν έδωσε ουσιαστικά ένα κακό παράδειγμα στον κύριο Μπέικερ, γιατί ο κύριος Μπέικερ επιθυμεί τώρα να δευτερολογήσει. Σας δίνω για δεύτερη φορά λοιπόν το λόγο κύριο Μπέικερ και συνέχεια στον κύριο Τόμας Μαν. Ε, um Ζητώ συγγνώμη, μία παρατήρηση ήθελα να κάνω. Προσέξαμε πως οι μεταφράσεις δημιούργησαν δυσκολίες και το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να δούμε πού οφείλεται αυτό. Δεν είναι βοηθάει και την εργασία μας. Euh, ευχαριστώ. Θεωρώ, θεωρώ πως με τη συζήτηση αυτή είχαμε ένα καλό παραδείγμα εργασίας του Κοινοβουλίου έλαβαν το λόγο οι σκιώδεις συγητές. Έχουμε και ένα γκρουπ επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Και το θέμα της επικοινωνίας, ο κύριος Μπέκερ είχε θέσει πολλά ερωτήματα για να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Επίσης μάλλον δεν το ξέρετε, μεταδιδόμαστε ζωντανά στο διαδίκτυο. Εάν κάποιος, λέμε, ήθελε να μας δει, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Οπότε το καλύτερο το οποίο έχω να πω στην Κομισιόν είναι καλό είναι να ε, κοιτάνε και το τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Και αυτό είναι κομμάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επίσης, ε, βλέπετε πως ε, δημιουργήσαμε εδώ πέρα την δυνατότητα από διαφορετικές θέσεις να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση η οποία είναι και ικανοποιητική και ε, επιτυχάνει πρόοδο. Να αναφερθώ σε κάτι σημαντικό που είπε ο κύριος Μπέκερ για δικαιώματα και ε, υποχρεώσεις. Πολλοί πολίτες δεν ξέρουν ε, τα δικαιώματά τους. Πώς θα έχουμε τότε ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, ευρωπαϊκή κοινή γνώμη όταν δεν ξέρουν ποιες δυνατότητες έχουν. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία για αυτό το θέμα. Το μήνυμα αυτό που θέλουμε να περάσουμε, πώς θα είναι ε, πιο λογικό και να λέμε στο τέλος πως πράγματι είναι καλή αυτή η ποικιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συμβιβασμοί αυτοί. Και όταν βλέπουμε πως έχουμε τόσες τροπολογίες, Είδαμε πως στο τέλος παρόλα αυτά είχαμε ε, κάποιο συμβασμό. Τώρα ανεξαρτήτως του εάν είναι ένα εκατομμύριο νομίζω επαρκεί. Την επόμενη φορά μπορούμε να πούμε πως πήγαν καλά τα πράγματα και θα έχουμε και άλλους φίλους στο πλευρό μας ε, και περισσότερη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ de formation. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, ζωντανά κιόλα. Κυρία Συγήτρια, έχετε τώρα το λόγο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας και να πω ότι θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει η αλλαγή που προτείνατε γιατί εν πάση περιπτώσει πέρα από αυτή την αλλαγή, πέρα από αυτή την αλλαγή έχει σημασία ποιο είναι το περιεχόμενο πίσω από αυτά τα λόγια. Δεν, δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι βρίσκεται πίσω από τις λέξεις. Είτε μιλήσουμε για πολίτες, είτε για ηθαγένεια ως προς τις πληροφορίες και το πώς θα προωθηθούν, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που έχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα ή θα έπρεπε να έχουν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν ή δεν έχουν γνώση αυτών των δικαιωμάτων. και γι' αυτό δεν θεωρούν ότι την χάνουν προστασίες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ε, προενεργή αντιμετώπιση έτσι ώστε αυτές οι ευάλωτες ομάδες να ενημερώνονται σε σχέση με τα δικαιώματά τους. Ε, ως προς την πρόταση της κυρίας Παπαδοπούλου, νομίζω ότι στην ε, Επιτροπή η Επιτροπή της Ουσίας θα πρέπει να αλλάξει τον ε, τίτλο για τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει δεν ε, υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν θα αντιταχθεί η Επιτροπή αν θέλετε να λάβουμε υπόψη το σκεπτικό του Φελίπε Γκονσάλες όταν είχε αρχίσει αυτή η καθαρά ευρωπαϊκή συζήτηση. Αυτή είναι η κληρονομιά του. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση αύριο και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα... και θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δίνω το λόγο στην κυρία Χάρκιν για το θέμα υπαριθμών 5 ως προς τη γνωμοδότηση για την αναγνώριση και προώθηση διασύνοριακών εθελοντικών δραστηριατήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο για να παρουσιάσει τις τροπολογίες συμβασμού. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για την πολύ καλή συνεργασία. Δεν υπάρχουν αντιγνωμίες. Ως προς τις τροπολογίες συμβασμού θα ήθελα να πω ότι ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών συνεισφέρει στο κείμενο και προσπαθώ να μην έχουμε επικαλύψεις, αλλά συμπεριλαμβάνω όλες τις βασικές ιδέες. Στην ε, μιλάμε για τον εθελοντισμό που δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικατάστατο της έμιστης εργασίας και επίσης πιστεύω ότι στην ΕΦ, ενώ ζητάμε από την Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες, ζητάμε να εστιάσουν την προσοχή στην επέκταση των ε, σχεδίων που προϋπάρχουν. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των εθελοντών. Στην H επίση είμαστε αναλογικοί. Λέμε στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για διασυνοριακά σχέδια, αλλά αυτό αφορά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν το ίδιο στα κράτη-μέλη. Και ως προς το I, μιλάμε για τη σύσταση ενός διασυνοριακού δικτύου οργανώσεων εθελοντών, και θα πρέπει να υπάρχουν νέα σημεία σύνδεσμοι εκεί που δεν υπάρχουν, σημεία επαφής, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ε, προϋπάρχουσες διαρθρώσεις. Ως προς τις μεμονωμένες τροπολογίες, όπως είπα, μερικές δεν μπορώ να τις δεχτώ, θα αναφερθώ σε μερικές. Και άλλες επειδή καλύπτονται από τους συμβιβασμούς. Ήρθα σε επαφή με την κυρία Ροντζίλη και μπορούμε να δεχτούμε δύο τροπολογίες με την προστίκη προφορικών. Ως προς άλλες τροπολογίες, οι 39 και 40 αναφέρονται στο διαβατήριο δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων. Δεν μπορώ να δεχτώ καμία από τις δύο, διότι δεν υπάρχει. Περιμένουμε η Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση και σε μία από τις τροπολογίες λέμε ότι θα έχουμε και την κάρτα εθελοντή, αλλά θα γίνει με την αντίστροφη σειρά. Αυτά θα γίνει με την αντίστροφη σειρά. Και επίσης ως προς την 52 δεν τη δέχομαι διότι λέει ότι προτείνει τη σύσταση ε, μίας, ενός πυρήνα εθελοντικών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Και νομίζω ότι θα το δεχτώ μόνο με προφορική. Αν συνάδελφοι έχουν άλλα σχόλια, ευχαρίστως να ε, επεκταθώ. Σας ευχαριστώ όμως γιατί δεν ήταν πολύ δύσκολη η εργασία μου. Ευχαριστούμε. Η κυρία ε, Ροντζούλη σε πρώτη φάση. Ε, εγώ... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για τη διαθεσιμότητά της στις προτάσεις συμβιβασμού. Αύριο θα ψηφίσουμε μία γνωμοδότηση για να δούμε κατά πόσο αναγνωρίζεται ο εθελοντισμός ε, και η αξία του γιατί 100 εκατομμύρια συμμετέχουν σε εθελοντική εργασία κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Πρόκειται για βασικές αρχές, ε, δικαιοσύνη, ηθαγένεια και ούτω καθεξής. Και αυτό υπογραμμίζεται. Το 2011 ήταν ένα πολύ, είχε ένα πολύ θετικό απολογισμό ως προς τον εθελοντισμό και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι ακριβώς μπορεί και πώς μπορεί να ανταποκριθεί η κοινωνία. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στους ευρωπαϊκούς στόχους όπως η κοινωνική συμμετοχή, η θαγένεια, εθελοντισμός, δικαιοσύνη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σαφές ε, νομικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό, διότι οι εθελοντές, μάλλον το καθεστώς των εθελοντών δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προσκόμματα. Θα υποστηρίξουμε τις 10 ε, τροπολογίες συμβασμού και όπως είπα στην εισηγήτρια, θα προτείνω στις, στις τροπολογίες 33 και 36 δύο προφορικές. Είμαστε θετικά διακείμενοι προς την γνωμοδότηση, αν και υπάρχουν ορισμένα σημεία διαφωνίας, γιατί ακούστηκαν επικρίσεις για το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δραστηριότητες εθελοντισμού οι οποίες θα μπορούσαν να εγγραφούν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο. Και νομίζω ότι μπορούμε διασυνοριακά να αναγνωρίσουμε την προσωπική πείρα του καθενός έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσα στα πλαίσια του θελοντισμού. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια. Η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εισηγήτρια η κυρία Χάρκιν είπε πως ε, ήταν δύσκολη η δουλειά τη Πράγματι, ειδικά αν σκεφτούμε την δημογραφική και την οικονομική κρίση, σημαίνουν πως η εθελοντική εργασία μπορεί εν μέρη να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά πρέπει βεβαίως να θυμόμαστε πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την, τον εθελοντισμό ως υποκατάστατο της εργασίας. Βεβαίω, οι εθελοντέ έχουν τι δικές τους ευθύνες, αλλά όταν μιλάμε για πραγματική δουλειά, πρέπει πάντα να προσλάβουμε κάποιον ο οποίος πληρώνεται. Δεν μπορούμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε την εθελοντική εργασία ως υποκατάστατο. Και βεβαίως η γύρανση του πληθυσμού σημαίνει πως θα χρειαστούν περισσότερους εθελοντές, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και έμπειροι και ειδικοί για να ασχοληθούν με τους ηλικιωμένους. Στηρίζουμε τους συμβιβασμούς και ίσως άξιζε να δούμε πώς θα μπορούσαμε τα ευρωπαϊκά αυτά έτη ε, με διάφορα θέματα να τα δούμε σε ένα σύνολο για να συνδέονται μεταξύ τους. Εν ολίγης, δεν είναι σωστό κατά την απόψή μου να ασχολούμαστε με ένα πρόβλημα μόνο για μία χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό φέτος που είναι το έτος ε, ε, ενεργού γύρανσης ε, να να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μια που σκεφτόμαστε λοιπόν τον εθελοντισμό, νομίζω πως ε, έχει μεγάλη σημασία και ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως πιο εύκολα αλλάζουν χώρα για να κάνουν και εθελοντική εργασία. Ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει να πάρει κανείς άλλο το λόγο, δίνω πάλι το λόγο στην συντάκτρια γνωμοδότησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνεται η ιδέα αυτή στις συμβαστικές τροπολογίες. Και λέμε επίσης και ποιε ικανότητες θα πρέπει να υπάρχουν επίσημες και ανεπίσημες στις 39 και 40, ιδίω στην τροπολογία 40, ως, μέλο, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Αυτού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων θα έχουμε και την ε, κάρτα αυτή θεροντισμού. Ουσιαστικά το αντίστροφο όμως θα πρέπει να συμβαίνει. Συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε από την προαλή σας, ότι θα πρέπει να διασυνδέσουμε κάπως τα θεματικά αυτά έτη και είχαμε και ένα θεματικό έτος για τη γύρανση, για το οποίο είχαμε διάφορες ε, πρωτοβουλίες στα πλαίσια του προγράμματος κομμήνιους. Θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν και τα προγράμματα αυτά, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους και για τον σχετικό με τους ηλικιωμένους εθελοντισμό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας. Σα ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τις τροπολογίες, τις συμβαστικές ε, αύριο. Κατά αυτόν τον τρόπο η ε, Επιτροπή Πολιτισμού θα λάβει υπόψη και τη δική μας την εργασία. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης, όπου βασιζόμαστε εδώ πέρα στην έκθεση της κυρίας Γιούτα Στάνρουκ όσον αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Εδώ θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με κάποιους προσκεκλημένους, ο οποίους δεν βλέπω ακόμα μέσα στην αίθουσα. Ας κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα προκειμένου να φτάσουν όλοι μας οι καλεσμένοι. Si chacun θέλει bien rejoindre θέση του, ότι θα μπορούμε... θέσεις για να ξεκινήσουμε πάλι τις si nos invités veulent bien και οι προσκεκλημένοι μας για να ξεκινήσει η ακρόαση. Μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις αυτές που λαμβάνουν χώρα για, την, για το μεγάλο αυτό νομοθετικό πακέτο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και έχουμε εκεί στο πλαίσιο αυτό ένα σημαντικό κείμενο για το οποίο είμαστε εμείς εισηγητές στην Επιτροπή μας και με την βοήθεια της συναδέλφου Γιούτα Στάινρουκ θα κάνουμε μια έκθεση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Δίνω καταρχάς, θα δώσουμε καταρχάς το λόγο στην εισηγητριά μας και στη συνέχεια ο καθένας από τους ομιλητές μας θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του προκειμένου να εκφράσει την τοποθέτηση αστικά της οργάνωσης που εκπροσωπεί. Κυρία Σιγήτρη, έχετε το λόγο. Äh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η σημερινή... Η σημερινή μήνυα ακρόαση μας δίνει την ε, ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να βοηθήσει και για την έκθεση που θα δώσω για μετάφραση την άλλη εβδομάδα. Ήδη συναντήθηκα δύο φορές με τους κοιόδης και ελπίζω να κάνουμε κάποια πράγματα προς σωστή κατεύθυνση και μια κοινή κατεύθυνση ε, για εκεί όπου βλέπουμε κάποια ανάγκη βελτίωσης των πραγμάτων Επίσης, διάσα πολλές φορές την πρόταση κανονισμού και δεν βλέπω εδώ πέρα ποια είναι η προστέμενη αξία της ε, σύμπτυξης των τριών προγραμμάτων Progress, Oires και μικροχρηματοδότησης, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς στόχους. Αντιλαμβάνομαι πως η Κομισιόν βεβαίως θέλει να απλοποιήσει τη δουλειά της, να μειωθεί το διοικητικό βάρος, αλλά εμείς δεν θα πρέπει να χάνουμε και την προσθέμενη αξία για τους πολίτες. Ήδη από τον τίτλο έχω σοβαρές αμφιβολίες. Η Κομισιόν ορίζει το πρόγραμμα αυτό για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία. Ε, τι κοινωνική αλλαγή μπορεί να ε, είναι προς το χειρότερο. Μπορεί να είναι προς το καλύτερο, πιο κοινωνική Ευρώπη, πιο πολλά δικαιώματα, αλλά μπορεί να σημαίνει και τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οπότε χρειαζόμαστε πρόγραμμα για την κοινωνική πρόοδο. Πρόσεξα πως η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ ασαφής σε πολλές περιπτώσεις και αφήνει πολύ μεγάλο χώρο στην Κομισιόν για να διαμορφώσει το πρόγραμμα. Προσπαθούμε λοιπόν να προσπαθώ να διαμορφώσω πιο το πρόγραμμα με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Καταπολέμηση της στόχιας, καλύτερες συνθήκες εργασίας, κοινωνική ένταξη. Αυτά δεν υπάρχουν κατά την άποψή μου εδώ πέρα και δεν υπάρχει εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, που είναι βασικό στατικό κομμάτι. Ναι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους των διαφόρων συμφερόντων με τις παρατηρήσεις τους να μας πούν τι θεωρούν, τι άποψη έχουν για τη δομή του προγράμματος, πού βλέπουν θεμενή αξία γιατί οι ειδικοί που ασχολούνται χρόνια με αυτό το θέμα ίσως να βλέπουν τα πράγματα και καλύτερα από μένα. Και θα ήθελα να ακούσω πώς εκτιμούν τα διάφορα υποπρογράμματα. Και μετά έχω και ερωτήσει μισό, αλλά αργότερα αυτό. Ε, Ωραία. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόνι ε, Ρόιτερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, κοινωνικής πλατφόρμας. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα λιγάκι. Καταρχήν ως προς τις γενικές παρατηρήσεις. Είναι ε, δύσκολο να βάζουμε μαζί πολλά προγράμματα διότι στο τέλος χάνουμε. Και είδαμε ότι πολλές φορές ε, είναι ικανοποιητικά όταν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε οργανώσεις που, εργάζονται, που ασχολούνται με αυτό το τομέα, διότι σήμερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται αυτή η συζήτηση. Ποιο είναι το νόημα του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου των πολιτών. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τάσσονται υπέρ του διαλόγου των πολιτών, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν οι οργανώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να δεσμεύονται και να καλύπτουν τα κενά που δεν καλύπτει η δημόσια διοίκηση ή που καλύπτουν κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Από πλευράς κοινωνικής πλατφόρμας καλύπτουμε 45 δίκτυα πλατφόρμες και αυτό που προσπαθούμε να καλύψουμε είναι ε, τις διάφορες οργανώσεις, έχουμε την Κόφασε, έχουμε πάρα πολλές οργανώσεις, την Σολιντάρ καταπολεμούν και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και επίσης έχουμε οργανώσεις οι οποίες παρέχουν ε, κοινωνικές υπηρεσίες, διότι χωρίς αυτές τις υποδομές δεν μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους της ε, Ευρώπης του 2020 από, το, από τότε που ίσχυσε αρχικά αυτό το πρόγραμμα βλέπουμε ότι έχουν επέλθει αλλαγές. Τώρα μιλώ πλέον για τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις αλλαγές που έχουν επέλθει έκτοτε και βεβαίως στην Ευρώπη του 2020. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την Ευρώπη του 2020 γιατί ε, δεσμευόμαστε, μιλούμε για αυτήν και σε ευρύτερο επίπεδο Μιλάμε για χρηματοοικονομική εξυγίανση και τίποτα άλλο. Για να κατανοήσουμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό και αυτή την εργασία θα πρέπει να ε, θυμόμαστε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω τις ε, κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας. Χρειαζόμαστε αυτά τα προγράμματα ακριβώς γι' αυτό γιατί υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη ανισότητα και η ίδια η Επιτροπή στην έκθεση της, του Δεκεμβρίου για την ανεργία και την κοινωνική ανάπτυξη μας έδωσε τα στοιχεία. Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας. Δείτε τα αριθμητικά στοιχεία καθεαυτά και θα δείτε τι ανισότητα υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όχι μόνο στις χώρες που ακολουθούν ένα πρόγραμμα λιτότητας. Αν ε, βάλουμε αυτά τα τρία σημεία μαζί, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πίσω από όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε σημασία και σε όλες αυτές τις ε, πτυχές. Από την πρόταση που έχουμε επιτάπητος θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ένα στεναρό χρηματοοικονομικό κανονισμό που, ο οποίος να καταπολεμά τις ε, κοινωνικές, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καταπολεμήσουμε καταρχήν την ανεργία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Νομίζω όμως ότι είναι για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό το ξέρουν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές υποδομές έτσι ώστε να ε, υπάρξουν και συνοδευτικά μέτρα. Προτείνουμε λοιπόν, όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική που είναι ένας γενικός ορισμός, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ερμηνείας, μετάφρασης και ερμηνείας, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική. Ίσως θα πρέπει να μιλάμε για κοινωνική προστασία και συμμετοχή. Επίσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτόν τον κύκλο ζωής του προγράμματος. Θα ήθελα να σας δώσω τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα για τη κοινωνική προστασία, την συμμετοχή και την καταπολέμηση της φτώχειας και την προτεραιότητα στην απασχόληση. Ξέρουμε ότι έχουμε 120 εκατομμύρια που βρίσκονται στο κατόφλι της ε, φτώχειας και γι' αυτό μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο ε, ακριβώς επιθυμεί να καταπολεμήσει την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και υπάρχει και η δέσμευση ε, του ποσού των 20 εκατομμυρίων, το οποίο είναι ευπρόσδεκτο κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης θα θέλαμε να μην υπάρχει γενική, αυτή η γενική μνήα της κοινωνικής πολιτικής, αλλά μιλάμε για κοινωνική συμμετοχή, προστασία και καταπολέμηση της φτώχειας. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος, αν συμπεριλάβουμε τα, τρίτα, τα τρία προγράμματα, να χάσουμε επί της ουσίας. Και νομίζω ότι τα προγενέστερα προγράμματα έδειξαν ότι επήλθε πρόοδος με βάση τις μη κυβερνητικές που συμμετείχαν σε αυτή την κοινωνική πλατφόρμα. Γιατί λοιπόν να μην την συνεχίσουμε. Το τρίτο σημείο, όπως είπα, αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Με το συνάδελφο από τα συνδικάτα ε, συναντηθήκαμε μπροστά στο κτίριο ε, Ζούστους Λήψιους για να συμμετάσχουμε στην μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνικός διάλογος και δεν θα πρέπει να μειωθεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό αυτό διάλογο. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ε, κοινωνικές οργανώσεις, ε, μη κυβερνητικέ και ούτω καθεξής. Έχει μεγάλη σημασία γιατί θα πρέπει να έχουμε τη σωστή διακυβέρνηση του προγράμματος, να μάθουμε ημέν από τους δε, να αντιλήσουμε διδάγματα και να δούμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για κοινωνική καινοτομία. Υπάρχουν γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κοινωνική καινοτομία, εξαιρετικά. Το πρώτο άκουσα το 86 στη Γαλλία και ακόμα καινοτομούμε. Έκτοτε καινοτομούμε. Βεβαίως υπάρχει και η ιδιαιτερότητα των ΜΚΟ και η καθημερινή τους εργασία. Θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς υπησέρχεται η διαφορά μεταξύ κοινωνικής ε, καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας, επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν με βάση αυτή την πύρα, τη συσσωρευμένη πύρα, να έχουμε διασαφηνίσεις. Επίσης όμως χρειάζεται χρηματοοικονομική υποστήριξη και αυτό αφορά τις οργανώσεις ε, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Δεν σημαίνει φιλανθρωπία, σημαίνει δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων εκεί όπου δεν παρεμβαίνει η δημόσια διοίκηση και να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν αυτό το κοινωνικό ρόλο ως ε, κοινωνικές μοικείο. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τον κοινωνικό διάλογο. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σε έναν ε, ε, σωστό, σε έναν σταθερό και στεναρό ε, χρηματοοικονομικό κανονισμό για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό ζητάμε να επέλθει κοινωνική αλλαγή. Γι' αυτό το πρόγραμμα της κοινωνικής αλλαγής και καινοτομίας 2014-2020, διότι μόνο έτσι θα καταπολύσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τα γενικά αυτά σχόλια που κάνετε, ενδεχομένω να δώσετε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις για τον απολογισμό της λειτουργίας ε, του προγράμματος Progress. Θα ήθελα τώρα για το τμήμα URES να δώσω το λόγο στην κυρία Κλοντ Ντενάκ Ντεργκάλ, η οποία εκπροσωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, για το ότι προσκαλέσατε την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για να μιλήσουμε για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόταση που μας εξέπληξε όπως και εσάς. Θα θέλαμε πραγματικά να γνωρίζουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της πρότασης. Είπατε ότι εντάσσεται στη γενικότερη νομοθετική πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο Περιμέναμε λοιπόν να λάβουμε κάποιες, περισσότερες, κάποιες περαιτέρω πληροφορίες μέχρι να παρουσιάσει το πρόγραμμά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλήρως την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό που θέλαμε να γνωρίσουμε είναι ποια είναι η χρήση που γίνεται εδώ πέρα των όρων καινοτομία και κοινωνική αλλαγή. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη κοινωνική καινοτομία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας απασχόλησε στα πλαίσια της ε, ΣΕΣ και χρησιμοποίησαμε και κάποιες ε, μελέτες που κάναμε το 2009 όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου κοινωνική καινοτομία, τι εμείς εννοούμε με τον όρο αυτό. Ανατρέξαμε λοιπόν στις μελέτες αυτές γιατί γίνονται διάφορες παράλληλες συζητήσεις με ορισμένους ε, καθηγητές πανεπιστημίου που ουσιαστικά θέλουν να εξαλείψουν εντελώς τον, την κοινωνική πρόοδο όπως αυτή έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια και σε μία τελευταία επαφή που είχαμε μεταξύ ΣΕΣ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είδαμε ότι ο επικεφαλής της τράπεζας αυτής μας είχε πει ότι έχει τελειώσει πλέον η περίοδος της περίφημης κοινωνικής προόδου. Όπως είπε και ο Κόνι Ρόιτερ, ο οποίος ήταν ε, μαζί μας στη διαδήλωση αυτή που έγινε στις Βρυξέλλες, αλλά και γενικά είναι παρόν σε όλες τις διαδηλώσεις που γίνονται στην Ευρώπη, πρέπει να επενθυμίσουμε τις βασικές μας αξίες και κάτι που βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά των προγραμμάτων, των διαφόρων δημοσιονομικών προγραμμάτων, είναι το ότι ακριβώς θα πρέπει να έχουμε αυτή την κοινωνική διάσταση. Και θα πρέπει για τα προγράμματα αυτά να έχουμε σαφώ, τα κοινωνικά προγράμματα να έχουμε σαφώς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ε, η αρχή της εταιρική σχέσης, όπως εμείς την καταλαβαίνουμε στα πλαίσια των ε, διαρθρωτικών ταμείων, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχυθεί. Κάθε φορά που μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κάθε φορά που μιλάμε για τον γενικό κανονισμό, θα υπάρχει δηλαδή ένα κώδικα συμπεριφορά ε, γι' αυτό. Πρέπει να ενισχυθούν λοιπόν οι σχετικέ διατάξει, οι σχετικέ προτάσει που συζητώνται τώρα στο Συμβούλιο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν προβλέπεται μια συγκεκριμένη εταιρική σχέση ούτε για το Progress ούτε για το Eures, μολονότι αναφερόμαστε ε, τουλάχιστον ευτυχώς στους κοινωνικούς εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή την βασική αρχή στην επεξεργασία του όλου αυτού προγράμματος, εφόσον το πρόγραμμα αυτό παραμείνει επιτάπητος. Και όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το Γιούρες θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια επιμέρους σημεία. Χάρη στην προηγούμενη θέση που είχα, ήμουνα σε θέση να παρακολουθήσω από το 1989 την πορεία του Γιούρες και τη διασυνοριακή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Και Στη συνεργασία που είχαμε τότε με τις επιχειρήσεις λέγαμε ότι θα πρέπει να υπήρχαν κάποια, α, κάποιες ευρωπαϊκές κοινωνικές διατάξεις που να ισχύουν στην νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του Γιούρες έχουμε τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και διασυνοριακά διαγραφεία προβλέπονταν συνολικά 21. Και έχουμε πέρα από τις δημόσιες αυτές υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι μολονό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί σαφώς υπέρ των υπηρεσιών αυτών, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και επομένως έχουμε και μια υποχώρηση των διασωνεριακών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων. και κατά αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί και η συμμετοχή σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Στις γενικότερες προτάσεις που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, γιατί το Euros αποτελεί ουσιαστικά μόνο ένα μέρος του προγράμματος, έχουμε ουσιαστικά δύο σημαντικές προτάσεις. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον θα πρέπει να προωθεί στην κινητικότητα και την απασχόληση, και προβλέπεται επίσης η ενίσχυση των δράσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Γιούρες από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και από τις διασυνοριακές εταιρικέ σχέσεις. Αυτό είναι θετικό για μας γιατί υπάρχει πάλι η έννοια της εταιρική σχέσης που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουμε και κάποιες επιτροπές παρακολούθησης, ε, υπάρχει και μια πιο αυτόματη συμμετοχή και θα ενισχυθεί και ο ρόλος των ε, περιφερειακών συμβούλων Γιούρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται από το 1994 για ζητήματα όπως η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία, τα δικαιώματα απασχόλησης, τα δικαιώματα των εργαζομένων οι οποίοι ε, εργάζονται σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εργασία τους. Είναι πολύ σημαντικό άλλωστε αυτό γιατί θέλουμε στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 να προωθήσουμε και την επαγγελματική κινητικότητα. Στα πλαίσια τώρα του συγκεκριμένου προγράμματος θα θέλαμε προφανώς να έχουμε τον άξονα γιούρες αλλά και να έχουμε και έναν κοινο, κοινοτικό συντονισμό δηλαδή να γίνουν κάποιες συντονισμένες συνεδριάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Τράπεζα Δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχουν και κάποια συντονισμένα προγράμματα κατάρτισης διαβίου μάθησης, τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται μέσω των συμβούλων στους οποίους αναφέρθηκα. Που χωλαίνει τώρα η πρόταση. Η διάρθρωση ανάμεσα στις δύο αυτές πτυχές, δηλαδή πώς θα εξελιχθούν στην πράξη τα πράγματα και ο προπολογισμό. Ξέρετε ότι είναι επίμαχο το σημείο αυτό. Ο προπολογισμό που χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συνολικό λοιπόν προπολογισμό, όλες οι σχετικές γραμμές προπολογισμού που εγκρίνονται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα χρησιμοποιηθούν εντελώ για τον ευρωπαϊκό αυτό συντονισμό. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Είναι εντελώς απαράδεκτο κάτι τέτοιο γιατί όπως σας είπα βλέπουμε ότι λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων κάποιες δραστηριότητες που προβλεπόντουσαν από τους κοινωνικούς εταίρους καταργούνται τώρα, ακυρώνονται στα πλαίσια της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτινόμενων προγραμμάτων. Τίθεται λοιπόν το σημαντικό αυτό ερώτημα. Τι ακριβώ πρόκειται να κάνουμε το ζήτημα του προπολογισμού. Θέλουμε προ αυτό κάποιε διευκρινήσει. Και επίση δεν θέλουμε όλο το δίκτυο Γιούρες, δηλαδή και το τμήμα του που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να ενταχθεί κατά αυτόν τον τρόπο στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προτιμούσαμε ανταυτού το δίκτυο Γιούρες να ενταχθεί ολόκληρο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει όμως να δημιουργηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός για να γίνει κάτι τέτοιο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί εξορίσμου να χρηματοδοτήσει κοινοτικά προγράμματα. Πρόκειται πάντως για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Είναι θεμελιώδες πάντως το πρόβλημα αυτό για μας και κατά την άποψή μας θα πρέπει να διατηρηθεί ο ρόλος της Γιούρες στις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. Δεν είναι μόνο το θέμα της απασχόλησης και των σχετικών συμβούλων και προτού να θεωρηθεί το δίκτυο EURES πριν το 2002 δηλαδή μια συγκεκριμένη αποστολή για το EURES ήταν η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου που μολονότι δεν προβλεπόταν στη συνέχεια στα νομοθετικά κείμενα, εμείς συνεχίσαμε τον κοινωνικό αυτό διάλογο, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν ιδιαίτερα θεμελιώδης όσον αφορά τις διασωνεριακές σχέσεις και ότι θα πρέπει να υπάρχει ο διάλογος αυτός με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης το δίκτυο EURES είναι, ανοίγεται όλο και περισσότερο προς τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Και αν δείτε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάμε απλώς για υπηρεσίες απασχόλησης, χωρίς να γίνεται καμία συγκεκριμένη μνήα στο αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Εμείς θέλουμε να διατηρηθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Δεν θα θέλαμε τα πράγματα να μην εξελιχθούν χωρίς κάποιον έλεγχο. Θέλουμε να υπάρχει η απαραίτητη πλαισίωση αν να χρησιμοποιήσουμε ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Αυτές οι παρατηρήσεις είχα να κάνω μέχρι στιγμής και συμφωνώ βέβαια και με τον προλήσασα, τον κύριο Κόνι Ρόιτερ, τον προλήσαντα με συγχωρείτε, ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα όσα ήδη έχουμε πετύχει στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και εμεί ως κοινωνικοί εταίροι, ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, βλέπαμε ότι δεν ήμασταν πλέον συνομιλητές όσον αφορά ζητήματα όπως η κατάρτιση, η κινητικότητα των εργαζομένων κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήταν ιδιαίτερα θετικό. Όσον αφορά τον τρίτο άξονα, αυτός δεν είναι δικός μου τομέας, αλλά συνδέουμε το Eures και με αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων. Αναφέρομαι στο Ζάσπερ, στο Τζέρεμι, στα προγράμματα αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εμπειρογνώμονες όμως μας λένε ότι τα προγράμματα αυτά ήταν ε, ιδιαίτερα βαριά, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών, ως προς την οργάνωσή τους, ως προς τη διάρθρωσή τους. Πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να αναλύσουμε ποια είναι η διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα τρία προγράμματα, στις τρεις αυτές ξεχωριστές πτυχές. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον, στον κύριο Ντανιέλ Σόροζαλ του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Μικροπιστώσεων, Μικροχρηματοδότησης. Για να τελειώσουμε με αυτό το γύρο, με αυτή την πρόταση τύπου marketing, σας δίνω το λόγο. Ο κύριος Μολινάρ δεν μπόρεσε να βρεθεί σήμερα μεταξύ μας. Έχετε εσείς το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος ε, του συναδέλφου που αρρώστησε και μου ζήτησε σήμερα το πρωί να τον αντικαταστήσω. Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω από τα σχόλια της συναδέλφου, να πω πως ε, μας μας ικανοποιεί η πρόταση. Δεν μπορώ να σχολιάσω για τη συμπληρωματικότητα και τα λοιπά στοιχεία, αλλά εάν ε, δούμε τους άξονες μικροχρηματοδότηση και κοινωνικών επιχειρήσεων όπου συνεργαστήκαμε στενά με την Κομισιόν είμαστε ικανοποιημένοι. Πρώτα απ' όλα καλωθορίζουμε την πιθανή επίπτωση στη δημιουργία θέσεων εργασία. Βεβαίω μιλάμε για επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχολούμενους αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είτε αναγκάζονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι λήψη άλλης εναλλακτική είτε γίνονται ένα υβριδικό είδος ε, υπαλλήλων που έχουν και μια δεύτερη δραστηριότητα ή άνθρωποι που είχαν στο παρελθόν ε, μισθωτή θέση εργασία αλλά τώρα αναγκάζονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Το προτινόμενο πρόγραμμα να αντιμετωπίζει δύο ζητήματα που μας ανησυχούσαν ιδιαίτερα. Αφενός την πρόσβαση στη χρηματοδότηση που στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος τομέας που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία ε, των ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι σημαντική η χρηματοδότηση αλλά και η πρόσβαση στην αγορά πρόσβαση σε δίκτυα κτλ. είναι εξίσου σημαντικά. Συγκεκριμένα τώρα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση θεωρούμε πως συνεχίζεται έτσι η γραμμή που είχε ξεκινήσει η Κομισιόν μέσω του μέσου μικροχρηματοδότησης για να υπάρχει μια πιο σταθερή χρηματοδοτική βάση για επιχειρηματίες. Όταν λέω επιχειρηματίες, μην σκέφτεστε μεγάλες ε, επιχειρήσεις, συχνά μιλάμε ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν άλλη λύση. Και θα ήθελα να προσθέσω επίσης το ότι πέρα από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται άλλες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι ε, καθοδήγηση, ανάπτυξης ε, των δραστηριοτήτων τους, που δεν είναι βεβαίως όπως η μικροχρηματοδότηση, αλλά είναι εξίσου σημαντικά για να επιτύχουν, γιατί μπορεί να ξεκινήσει κανείς μια νέα επιχείρηση αύριο μέσω ενός δανείου που έλαβε χτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ε, θα μπορέσει να καλύψει τις δραστηριότητες των πρώτων ετών χωρίς επιπλέον στήριξη. Οπότε πρέπει να ενισχυθούν συνέργειες, συντονισμός με τους υφιστάμενους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ειδικά στο εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε οποιοδήποτε νέος επιχειρηματίας να έχει πρόσβαση όχι μόνο στη χρηματοδότηση, για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ε, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν η πρόταση περιλαμβάνει μία απέτηση για οποιονδήποτε συμμετέχει στο πρόγραμμα. Γιατί όπως είπαμε είναι πράγματα που χρειάζονται και παίζουν κρίσιμο ρόλο. Ε, όταν βεβαίως εκπροσωπώ το δίκτυο ευρωπαϊκής μικροχρηματοδότησης, συμπεριλαμβάνει αφενός ΜΚΟ, τράπεζες, ε, αποταμιευτικούς συνεταιρισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν είναι τράπεζες. Το βασικό κοινό του σημείο είναι πως συνεργάζονται με ευπαθείς ομάδες και κατά κανόνα δεν καλύπτονται ε, αυτές οι ομάδες από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα για λόγους πιστοληπτικής ικανότητας ε, κτλ. Οπότε καλωσορίζουμε τον άξονα αυτό, ο οποίος ε, δίνει μία πιο αηφόρο χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμα, αλλά επίσης αντιμετωπίζει και το ζήτημα της οικονόμησης δυνατοτήτων των παρόχων μικροχρηματοδότησης. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ και καιρό και παρά το ότι κάποια προγράμματα υπήρχαν μέσω διαφόρων μέσων, θεωρούσαμε πως ε, μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και ο λόγος για την αύξηση αυτής της ε, θεσμικής ικανότητας είναι ότι αφενός βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για αυτή τη χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων και αφετέρου οι οργανώσεις που εκπροσωπώ δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την ζήτηση γιατί δεν έχουν οριμάσει αρκετά σε περισσότερε περιπτώσει λειτουργούν εδώ και 10 χρόνια και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζήτηση. Οπότε το ζήτημα αυτό έχει κρίσιμη σημασία. Θα ήθελα να προσθέσω πως το προτινόμενο μέσο έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Πως ε, υπάρχει μια κεντρική διαχείριση. Μέχρι τώρα είχαμε τρεις-τέσσερις ε, γενικές ε, διευθύνσεις και θα, καλό θα ήταν να απευθυνόμαστε σε έναν μόνο. Και για τη χρηματοδότηση, την ε, αύξηση των δυνατοτήτων, τεχνική αρρωγή κτλ. Δεν ξέρω αν ο συνδυασμό αυτών των αξώνων με τα άλλα δύο μέρη του προγράμματο είναι επιθυμητό ε, από μια πιο συνολική σκοπιά, αλλά εμεί θεωρούμε πω οι συνέργειες είναι σημαντικέ και βεβαίω καλωσορίζουμε το ότι είναι ένα μέρο ενό ευρύτερου προγράμματος. Γιατί η μικροχρηματοδότηση συνήθω είναι κάτι το οποίο θυμάται κανείς εκ των υστέρων και δεν είναι ούτε ακριβώς ε, θέμα τη χρηματοδότηση ούτε κοινωνικό ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να αποδώσει. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε αυτές τις συνοδευτικές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για του μικροεπιχειρηματίε και του νέου επιχειρηματίε γενικώ. Θεωρούμε πως μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για να διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία μεταξύ ε, οργανισμών μικροκληματοδότησης και παρόχων ε, υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων. Κάπως λοιπόν πρέπει να τονίσουμε το θέμα αυτό και οπωσδήποτε η κεντρική διαχείριση μπορεί να βοηθήσει αυτό. Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε στη συμπληρωματικότητα με τις κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι κάτι το νέο ακόμα ως ιδέα και θα θέλαμε να έχουμε παρόμοια πράγματα, ομοειδή πράγματα μαζί γιατί βεβαίως ε, μπορούμε να το δούμε αυτό ή μικροεπιχειρήσεις και μικροχρηματοδότηση να το δούμε πως, ε, ως ένα είδος ε, κοινωνικής έτσι, πολιτικής μπορεί να θεωρήσει κανείς υποδείγματα ή κοινωνικές επιχειρήσεις και βεβαίω μπορεί να χρηματοδοθεί ένα καινοτόμο επιχειρηματία με μια νέα ιδέα που μπορεί αργότερα να γίνει κοινωνική επιχείρηση αλλά θα πρέπει να πάει από του κατάλληλου τους χρηματοδότηση. Το ζήτημα βασικά είναι πως ε, δεν έχουν τη δυνατότητα οι εταιρείε αυτέ να ασχοληθούν με μεγαλύτερους οργανισμούς. Οπότε πρέπει να παραμείνουν χωριστά αυτά τα πράγματα. Οπότε βασικά από την δική μας τη σκοπιά θα θέλαμε να τονίσουμε τη στήριξή μας στον άξονα της κοινωνικής αλλαγής γιατί βεβαίως αφορά δύο ζητήματα που μας απασχολούν εδώ και καιρό δηλαδή μια σταθερή πηγή μικροχρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία στο μέλλον στην Ευρώπη και βεβαίω η αύξηση των δυνατοτήτων τους για να γίνουν και πιο όριμες αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουμε επίσης κάποιες παρατηρήσεις επί των λεπτομεριών. Εάν δείτε τον προϋπολογισμό που προτείνεται, 184 εκατομμύρια πάνε στην μικροχρηματοδότηση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, από τα οποία 80 εκατομμύρια πάνε στη μικροχρηματοδότηση. Το ποσό αυτό θα μοχλευθεί μέχρι και στο πλάσιο και φτάσει τα 500 εκατομμύρια. Αν δούμε δε την υφιστάμενη εμπειρία, ε, είναι λίγο φιλόδοξο αυτό το νούμερο. Δύο-τρεις φορές η μόχλευση είναι λογικό. Οπότε μιλάμε για 8 εκατομμύρια μετά που πάνε στην αύξηση των δυνατοτήτων των ε, διαφόρων της οργάνων και ε, δεδομένου του ότι θα στηριχθούν 80 τέτοιοι οργανισμοί, το ποσό, ποσό αυτό είναι χαμηλό. Ίσως 20 με 30 τέτοιες οργανώσεις θα μπορούσαμε να στηρίξουμε, αλλά ίσως αυτό θα το δούμε μετά στις λεπτομέρειες. Ο στόχος των 50.000 μικροδανείων είναι επισημαντικός. Είναι ένα στόχος όχι ιδιαίτερα φιλόδοξος, μιλάμε για ένα 10% αύξηση του ποσού που δίνεται αυτή τη στιγμή Επίσης Μπορούσε λοιπόν να είναι και πιο φιλόδοξος στόχος. Και Γενικώ θα θέλαμε ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με τα υπόλοιπα του προγράμματος να πούμε πως καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση ε, για μικροχρηματοδότηση και από τη σκοπιά μας θεωρούμε πως αντιμετωπίζεται στις ανάγκες του, του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Merci, je vais donc maintenant euh, συζήτηση. Και δίνω το λόγο στην κυρία Μωρά Σαρτιά και μετά στην κυρία Κίνκα Κόνς. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ και τους προσκαλεσμένους μας. Το πρώτο θέμα αφορά το ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση της κρίσης για την επόμενη φάση των προγραμμάτων. Και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στους παρεμβαίνοντες. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, συμφωνούμε όλοι ως προς τους πολιτικούς στόχους, όπως έχουν προσδιοριστεί δηλαδή επαγγελματική συμμετοχή και ενσωμάτωση, καταπολέμηση και καταπολέμηση της φτώχειας. Έτσι ώστε να έχουμε συμφωνήσει επ' αυτού για να απαντήσουμε στο δεύτερο σκέλος. Η κοινωνική εταιρική σχέση υπερτονίζεται και, εν πάση περιπτώσει, ορίζεται μέχρι πού θέλουμε να προχωρήσουμε στον ορισμό της κοινωνικής εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς επ' αυτού και θα πρέπει να εργαστούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, να γίνει ένας διάλογος με τα κράτη, μέχρι πού θέλουμε να προχωρήσουμε. Εάν προχωρήσουμε πολύ μακριά δεν θα μπορούσαμε να προσκρούσουμε σε δυσκολίες. Δεν θα πρέπει να είμαστε κάπως ευέλικτοι. Και τέλος, δεν θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ μεθόδου, μεθοδολογίας, μεθοδολογίας εργασίας για να ακολουθήσουμε μία τακτική κανονική διαδικασία, αν και όρος δεν σημαίνει πια τίποτα, και να υπάρχει μία κινητοποίηση ως προς τα προγράμματα. Διότι πέρα από τη μάχη των αριθμών, έχει σημασία η μάχη της κινητοποίησης πώς μπορείτε να περάσετε σε μία μέθοδο κοινωνικής εταιρικής σχέσης στην κινητοποίηση καθε αυτή και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Τέλος, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ίσως υποτιμήσαμε κάπως. Αφορά την κατάρτιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς ε, αυτή την κινητοποίηση. Και τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω, γιατί δεν το θίξατε εσείς, σε αυτή τη νέα στρατηγική θέλουμε μέτρα αντικτύπου, γιατί όλοι βρίσκουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύστοκη αυτή η έλεγχη πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αποτιμήσουμε την ευρωπαϊκή κινητοποίηση με στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Kinga Guns. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο και μία ερώτηση. τους εμπειρογνώμονες συμφωνώ ότι όταν μιλάμε για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία είναι κάτι το πολύ ωραίο αλλά πρόκειται για τα προγράμματα, τα τρία προγράμματα που είχαμε κατά την ε, προηγούμενη περίοδο. Δεν βλέπω και τόσο μεγάλη καινοτομία. Καθίσταται όμως σαφές ε, ένα είδος καινοτομίας ότι υπάρχουν λιγότεροι πόροι από ό,τι στο παρελθόν. για το μέσο μικροχρηματοδότησης, για το γιούρες. Θα πρέπει αυτά να ενταχθούν σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μία άλλη πλαισίωση, στα πλαίσια του ΕΚΤ. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό κατά πόσο είναι η σωστή λύση, γιατί μιλάμε για διαφορετικά προγράμματα, δηλαδή διατροφικής ε, βοήθειας και ούτω καθεξής. Ως ως προς το μέσο μικροχρηματοδότησης, παρακολουθώντας το πρόγραμμα εξ αρχής, διαπιστώνω ότι αναπτύσσεται διαφορετικά στις διάφορες χώρες και αυτό αφορά και τον κανονισμό, το, το, περιθώριο ρύθμισης μάλλον στις ε, διάφορες χώρες. Ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό τον κανονισμό ή αυτούς τους κανονισμούς έτσι ώστε να είναι πιο προσπελάσιμη για τους ενδυνάμει χρήστες. Ανάλογα με το ιστορικό της μικροχρηματοδότησης διάφορες χώρες. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για πόρους, αν επαρκούν ή όχι γιατί δεν λαμβάνουμε και το στοιχείο όχι μόνο της ρύθμισης αλλά και της γενικότερης ε, νουθεσίας και τους ενδυνάμει πελάτες, τους ενδυνάμει χρήστες. Βλέπετε αυτή την πτυχή ε, αυτής της ρύθμισης ή του κανονισμού μικροχρηματοδότησης. ένα σχετικά καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέεται με την ε, μικροχρηματοδότηση αφορά τις επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να ε, οδηγήσουν σε δανειοδοτήσεις στους μικροεπιχειρηματίες ή φορείς. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πραγματικά καινοτόμες αλλά δεν είναι προσβάσιμες σε όλους. ιδιαίτερα ως προς τις τρίτες χώρες. Πώς φαντάζεστε αυτές τις ρυθμιστικές αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του μέσου μικροχρηματοδότησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέεται βεβαίως και με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω και το χρόνο που περνάει και αρχίζω και ανησυχώ. Θα ζητήσω λοιπόν από τους ομιλητές μας να μιλήσουν σύντομα. Θα περιοριστώ σε τρία σύντομα πραγματάκια. Ε, για τους ειδικούς μας. Κυρία Στάινλουκ ήδη μας είπε πως έχουμε ήδη εργαστεί. Υπάρχει μια πρόταση της εισηγήτριας να πούμε πως ναι θα θέλαμε να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες κάτω το οποίο σημαίνει πως η Κομισιόν μετά δεν θα είναι μόνη της αλλά υπάρχει διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έχουμε Άρα, μια οργάνωση ομπρέλα των δικαιούχων του προγράμματος που θα είναι σε μια επιτροπή παρακολούθησης και διοίκησης στην εφαρμογή και τον έλεγχο. Και βεβαίως θα μπορούν να ε, προχωρήσουν στην ε, στην αυτών των προγραμμάτων. εξαρτώσει, δηλαδή των στόχων αυτού του προγράμματος, θα μπορούν να ασχολούνται με τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Ποια είναι η θέση σας από αυτού. Δεύτερον, η πρόταση των συνδικάτων το EURES να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί η δουλειά του EURES ε, όσον αφορά και την πλατφόρμα αλλά και τις ε, διασυνοριακές εταιρικέ σχέσεις είναι μια ευρωπαϊκή δουλειά και νομίζουμε άρα πως ε, δεν είναι εθνική υπόθεση. Το Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο εφαρμόζεται εθνικά. Τρίτον, το αποθεματικό, το αποθεματικό το αφήσαμε. Και Βεβαίω μιλάμε για το ότι πρέπει σε ορισμένε περιπτώσει να γίνουν καινοτόμοι διαγωνισμοί για τα πιλωτικά έργα. Θα με ενδιέφερε λοιπόν εδώ πέρα να γνωρίζω σε ποιο βαθμό οι εταίροι συμφωνούν με τέτοια πιλωτικά έργα τα οποία θα ξεκινήσουν και τα οποία θα συλλέξουν σε εθνικό επίπεδο τις καλύτερες εμπειρίες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δηλαδή υπάρχουν πιλωτικά έργα τα οποία θα εκτελεστούν, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αφήνουμε μετά ανοιχτή την δυνατότητα μιας επιτυχού ε, εφαρμογής ε, να έχουμε, δηλαδή ένα μέσο το οποίο θα μπορεί να αντιδρά και ποια είναι η δυνατότητα αντίδρασης στην κρίση που δεν υπήρχε στο παρελθόν και ποιες είναι οι αναγκαίες δράσεις από πλευράς Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρκιν και Ντέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί έχουν απαντηθεί ήδη κάποιες από τις ερωτήσεις μου. Ασχοληθήκαμε ήδη με το ζήτημα της συμμετοχής, της συμμετοχής δηλαδή των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών. Το δικό μου το ερώτημα ομοιάζει με αυτό που ακούστηκε. Ποια είναι η δική σας η άποψη, δεύτερον, όσον αφορά την μικροχρηματοδότηση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να δούμε ποια είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο και είχαμε δύο πολύ καλές συναντήσεις μέχρι στιγμής. Να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Πώς βλέπετε εσείς τη διαφορά αυτή. Πιστεύετε ότι αλληλοσυμπληρώνονται ή ότι ενδεχομένω να πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να ισχύουν ξεχωριστοί κανόνε, αλλά έστω ξεχωριστοί μηχανισμοί. Αναφερθήκατε επίση στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των παρόχων μικροχρηματοδότηση. Νομίζω ότι Τζέρεμ είναι το πρόγραμμα αυτό, έτσι δεν είναι θα μου πείτε τέλο πάντων ποιο είναι το αρμόδιο πρόγραμμα. Σύμφωνο πάντως ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτή τη δημιουργία ικανοτήτων. Αναφερθήκατε στον στόχο των 50.000 μικροχρηματοδοτήσεων, δανείων μικροχρηματοδότησης. Ποιος πιστεύω ότι θα ήταν ασφιλόδοξο στόχος. Και όσον αφορά τώρα τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επέλθουν, ποιες αλλαγές θα προτείνετε για τους τρεις αυτούς άξονες. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελή και ο κύριος Μπουλόν στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχάς για την προκαταρκτική ευθεργασία που έχει κάνει. Συμφωνώ σε έναν βαθμό με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Δεν είναι φυσιολογικό το δεν έχουμε ακόμα αξιολόγηση. Έχουμε, λάβαμε σήμερα την αξιολόγηση του Progress, 300 σελίδες, ενώ δεν υπάρχει αξιολόγηση για τα άλλα προγράμματα. Και δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να προετοιμάσουμε σωστά την εργασία μας. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπαν από την κοινωνική πλατφόρμα. Μην ξεχνάμε και τη φτώχεια η απασχόληση δεν είναι το μέσο το οποίο μόνο του θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φτώχειας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι τι εννοείται με την ε, κοινωνική καινοτομία, δηλαδή ποια θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Γιατί επί του παρόντος βλέπουμε ότι όλοι μιλάνε για κοινωνική καινοτομία. Τι ακριβώς εννοούμε. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει η κοινωνική οικονομία να ενταχθεί στην μικροχρηματοδότηση. Στο κείμενο όμως λέγεται κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, εσείς που γνωρίζετε τον τομέα και τους μηχανισμούς αυτούς, τι καταλαβαίνετε από τη φράση αυτή. Αυτά είχα να σας πω. Τις τρεις αυτές ερωτήσεις έκανα. Ο κύριος Μπουλό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, παρεμβαίνοντες euh, και τους σκιώθους. Και ως προς τις παρεμβάσεις, τις ζωηρές παρεμβάσεις που έγιναν, θα ήθελα να πω ότι η απασχόληση δεν είναι ο μόνος ε, τρόπος να φτάσουμε στους στόχους 2020. Υπάρχουν πολλά δίκτυα ε, στην περιφέρεια της απασχόλησης, στο τομέα της στέγασης, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και ούτω καθεξής. Υπάρχουν οι ΜΚΟ, οι κοινωνικοί εταίροι και η επιτόπια δράση. Πώς ορίζεται αυτή την εταιρική σχέση σε τοπικό επίπεδο ως προς τη χρηματοδότηση θα ήθελα να πω ότι ως προς τις ε, γενικές κατευθύνσεις συμφωνώ και ιδιαίτερα ως προς την τοπική διάσταση του θέματος της απασχόλησης, να υπάρχει κινητικότητα κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε διασυνοριακό επίπεδο. Για τη μικροχρηματοδότηση πιστεύω ότι αποτελεί προτεραιότητα. Η ΜΜΕ θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του σκεπτικού μας, διότι πολλοί δεν έχουν πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και αυτή η πλατφόρμα καινοτομίας που δεν είναι απόλυτα σαφής θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να δούμε τι είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κοινωνικά υπεύθυνες, ποια είναι τα οικονομικά τους αποτελέσματα τη στιγμή που έχουν ε, που καλύπτουν και αυτό το καθαρά ε, κοινωνικό σκεπτικό. Ως προς την καινοτομία, δεν μπορούμε να μιλάμε για ομαδοποίηση ή συγχώνευση αυτών των προγραμμάτων επιδοτήσεων θα πρέπει να ορίσουμε την ενία θηρίδα, τα προγράμματα, το ΕΚΤ και θα πρέπει να άρουμε τα προσκόμματα που υπάρχουν στην κοινή μας στην ενία αγορά ως προς την αποτίμηση Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ευεργετηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στα πλαίσια της μικροχρηματοδότησης. Τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές εικόνες για τους δικαιούχους. Πώς κρίνετε αυτή την αξιολόγηση και τέλος Ακόμα κι αν ε, εξαρτώμεθα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, μιλάμε και για το Ταμείο Συνοχής και δεν ξέρω κατά πόσο μέσω αυτής της ε, έκθεσης θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί. Η συγγήτρια θα ήθελε κάτι να μας πει. Ναι. Ευχαριστώ. Τα ερωτήματα που ακούστηκαν νομίζω οδηγούν και σε αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει. Έχω κάποια ερωτήματα για το θέμα ε, διακριτική μεταχείριση και ισότητα. δεν ήταν, ε, δεν ε, ήταν πριν στο Progress και έχει φύγει. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι γιατί έγινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεύτερο ερώτημα, τι ήταν στο παλαιό Progress μέσα, τι λείπει τώρα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν πρέπει να χαθεί ε, με κανένα τρόπο. Στον κύριο Σόκοσάλ η απάντηση στο υποπρόγραμμα, η απέτηση στο υποπρόγραμμα για κοινωνικέ ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσει γιατί η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι συγκεκριμένη. Πώς βλέπετε κάποιο ύψος ε, γραμμών πιστώσεων που δεν, ε, δεν θα υπαρκούσαν. Πώς θα να διαμορφωθούν. Αυτές είναι οι πρώτες μου ερωτήσεις. Ας δώσω το λόγο με την αντίστροφη σειρά. Δανιέλ Σοροσάλα, για πέντε λεπτά. Πολλά θέματα ως προς τον κανονισμό, το θέμα της μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει εναρμόνιση και αν δούμε τις διάφορες οργανώσεις, τις χώρες έχουν διαφορετικό καθεστώς, υπάγονται στα Υπουργεία, ε, μερικές είναι ΜΚΟ, άλλες εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες, α, ε, για άλλες δεν υπάρχει απόλυτη ρύθμιση, γι' αυτό σίγουρα θα ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός. Να ε, αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των οργανώσεων έτσι ώστε να έχουμε έναν εναρμονισμένο κανονισμό. Ποια στοιχεία μπορούμε να έχουμε, αριθμητικά στοιχεία, ποια είναι η στοχοθέτηση, ποιοι είναι οι πελάτες και πώς θα, γίνονται, πώς θα γίνεται η κατανομή των κονδυλίων. Βεβαίως η ρύθμιση είναι κάτι το δύσκολο, διότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε, να μειώσουμε τη δυνατότητα καινοτομία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκόμματα του τομέα. Ως προς τις νέες πρωτοβουλίες, ε, μεταξύ ομοτήμων θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Θα πρέπει να δούμε ενδυνάμει σχέδια με ενδυνάμει χρηματοδότες. Αυτό μπορεί να γίνει με κοινωνικά μέσα, αλλά δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτό το παζλ δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε τις ψηφίδες. Είναι μια δυνατότητα την οποία θα προωθήσουμε. Και βεβαίως αφορά και την ατζέντα κοινωνικής καινοτομίας. Θα πειραματιστούμε. Δεν ξέρουμε. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η αποκοινού χρηματοδότηση θα βοηθούσε και θα απελευθερώσει τα κονδύλια και τους πόρους έτσι ώστε να έχουμε μια λιγότερο παραδοσιακή προσέγγιση ως προς την ε, Επιτροπή Διευθυντήριο ε, για να μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές θα είμαστε υπέρ αυτής, θα την προωθήσουμε ως προς τον συμπληρωματικό χαρακτήρα και την εταιρική σχέση, την κοινωνική εταιρικότητα. Υπάρχουν ε, τρεις βασικές ιδέες. Η μικροχρηματοδότηση και ο επιχειρηματικός χαρακτήρας, η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το διαφορετικό. Μιλάμε ότι ε, χρηματοδοτούμε μικρές επιχειρήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά ε, χρηματοδοτούμε οργανώς. Δηλαδή το ένα σκέλος χρηματοδοτεί ανθρώπους, το άλλο επιχειρήσει. Υπάρχουν και κοινά, δηλαδή κάποιος... Ε, με νέες ιδέες θα μπορούσε να ζητήσει ε, πόρους από τη μικροχρηματοδότηση. Μετά όμως θα μπουν στη, όλα αυτά θα μπουν στην εντολή της μικροχρηματοδότησης. Δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο αυτή η καινοτόμος ιδέα θα μπορούσε να παραμείνει εκεί όταν υπάρχει ευρύτερη εμβέλεια. Μπάς περιπτώσει αυτό είναι το σημείο κίνησης Άρα η, μικροχρηματοδότηση μπορεί να χρηματοδοτήσει φυσικά πρόσωπα αλλά και οργανώσεις. Μετά περνάμε αλλού. Ως προς την κοινωνική εταιρικότητα πρόκειται για μία νέα έννοια και για εμάς. Θεωρούμε ότι τα κοινωνικά θέματα θα πρέπει να τα βλέπουμε μέσω επιχειρηματικότητας και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλουμε κάτω από, από το ίδιο φάσμα. Επειδή έχω ε, δουλέψει σε ΜΚΟ, θεωρούμε ότι ορίζουμε νέες εντολές και πολλές φορές μιλάμε για πόρους που δημιουργούμε εμείς και προωθούμε εμείς, άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ε, κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό σχέδιο, αλλά ε, ενέχει μία δυναμική και μιλάμε για πόρους οι οποίοι δεν είναι πάντα διαθέσιμοι. Αν πάω σε μια τράπεζα και θέλω να χρηματοδοτήσω ένα μηχανισμό για να ασχοληθώ με τον κοινωνικό αντίκτυπο των επενδυτικών ταμείων, για τα παιδιά και την εκπαίδευση. Δεν θα, ξέ, δεν θα ήξερα ποιο είναι το σημείο εκκίνησης. Είναι όμως ένα ε, θέμα που αφορά τον οικονομικό τομέα, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει ένα κοινωνικό ζήτημα. Για να δούμε πώς ε, ορίζεται αυτός ο αντίκτυπος. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς όπου θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα για να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα. Είναι κάτι το νέο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το υποτιμήσουμε, γιατί και η μικροχρηματοδότηση κάποτε ήταν κάτι το καινούριο. Δεν, ε, δεν ήταν ε, παρακάτι το καινοτόμο για κάποιον που δεν είχε τραπεζικά εχέγγυα. Ως προς την πρόσβαση τους τύπους πρόσβασης. Νομίζω ότι το προανέφερα για την ε, δυνατότητα ε, οικοδόμησης και προώθησης σχεδίων μέσα στα πλαίσια ε, οργανώσεων. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τους πόρους για την επιχειρηματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δεν ε, εργαζόμαστε επ' αυτού, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένας ε, τρόπος ε, ένα σημείο ανάπτυξης και ως προς την αξιολόγηση είναι πάρα είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις των προγραμμάτων μικροχρηματοδότησης, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν τρία θέματα που μπορούμε να αποτιμήσουμε, πόσες επιχειρήσεις, πόσες θέσεις εργασίας και κατά πόσο είναι βιώσιμες. Και να δούμε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις και αυτές τις θέσεις. Αυτά τα ολίγα σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντενάγκτερτάρλ εκπροσωπώντας την ΕΣΕΣ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες αυτές στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω μπροστά μου. Θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία ορισμός της κοινωνικής καινοτομία, εταιρικές σχέσεις και γιούρες. Όσον αφορά το πρώτο, ορισμός για την κοινωνική καινοτομία. Εμείς ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μια κοινωνική οπισθοδρόμηση. Δεν θέλουμε να τελειώσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ξέρουμε όμως και τι θέλουμε να πετύχουμε. Για παράδειγμα και σε σχέση με την κοινωνική καινοτομία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμα και για κοινωνική αιρεσιμότητα. Δηλαδή μιλάμε πολύ συχνά για μακροοικονομική αιρεσιμότητα για την πολιτική συνοχή. Εμείς θα ζητήσουμε να υπάρξει και μία κοινωνική αιρεσιμότητα, κοινωνικές προϋποθέσεις δηλαδή, να τηρείται η ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία και θα ζητήσουμε επιπλέον και την χρησιμοποίηση των προγραμμάτων αυτών για να υλοποιηθεί η κοινωνική ατζέντα, για την οποία μιλάμε πολύ λίγο και στο παρελθόν την ονομάζαμε μια ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Οι ιδέες υπάρχουν. Και αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια συνεκτικότητα, να συνδυάζεται το πρόγραμμα αυτό με άλλα προγράμματα, με άλλους φορείς και με τους σχετικούς προπολογισμούς που έχουμε, τους επιμέρους, στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουμε μια προσέγγιση κάπως ασαφή όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, με πολλούς διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εστιάσουμε καλύτερα και ευτυχώ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει την απαραίτητη αυτή εργασία. Και στα πλαίσια της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες. Αν δεν δείξουμε όμως την απαραίτητη προσοχή, νομίζω ότι θα αναλωθούμε τόσο πολύ σε τόσες διαφορετικές συζητήσεις που τελικά θα χάσουμε και την ίδια την ουσία. Δεν θα υπάρχει ένα πραγματικό περιεχόμενο στον όρο κοινωνική πολιτική. Να αναφερθώ και λίγο στις εταιρικές σχέσεις. Και ξέρετε ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Και ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κοινωνικής ένταξης. Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της απασχόλησης, αλλά επιτυγχάνεται τελικά κυρίως μέσω της απασχόλησης. Δείτε τι γίνεται στις κοινωνίες μας. Αν δεν έχουμε θέση απασχόλησης, αν δεν έχουμε δουλειά και μάλιστα ποιοτική δουλειά, δεν καταφέρνουμε να ενταχθούμε και κοινωνικά. Εμείς δίνουμε τεράστια μάχη προκειμένου να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τις επισφαλείς θέσεις εργασίας. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίζουμε να προωθούμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εργάζονται για το στόχο αυτό. Επιθυμούμε να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση των ανθρώπων και θα ήθελα κατά αυτόν τον τρόπο να αφαιρθώ και σε ένα βασικό στόχο της στρατηγικής 2020, να μειωθεί ο αριθμός των φτωχών ή τουλάχιστον να μειωθεί το ποσοστό των φτωχών στις κοινωνίες μας. Και για να βιτευτεί κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό τη εταιρική σχέση, ακόμα και την εταιρική σχέση που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Όταν λέμε εταιρική σχέση, ουσιαστικά τι εννοούμε, τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εταίροι, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένου κανόνε, οι οποίοι υφίστανται ήδη στα πλαίσια των διαφορετικών ταμείων, αλλά δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε ένα σαφή ορισμό και σαφείς πρακτικές οι οποίες να είναι πανομοιότυπες σε όλες τις χώρες και χρειαζόμαστε και ένα σαφή ορισμό για το ρόλο που θα πρέπει να δραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Αναφέρομαι επίσης και στο ρόλο που θα πρέπει να δραματίσουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Και στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους εταίρους και βέβαια οι κύριοι συνομιλητέ είναι οι κοινωνικοί εταίροι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ε, αποκλείουμε όλο και περισσότερο τους κοινωνικούς εταίρους και αποκλείουμε και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και αυτό σχετίζεται και με την όλη κατάσταση της οικονομικής κρίσης που γνωρίζουμε, των προγραμμάτων λιτότητας. Ας δούμε τι έγινε στο Βέλγιο αυτή την εβδομάδα. υπήρχαν, έγινε μια έντονη διαδήλωση εργαζομένων που ήρθαν από τη Γερμανία για μια εταιρεία η οποία πρόκειται να μετατοπίσει της, την παραγωγή της και ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να πάρουν την, τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν στην εταιρεία αυτή. Και αυτό χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτο, αλλά καταλήγουμε σε τέτοιες καταστάσεις τελικά. Αν δεν προασπιζόμαστε σωστά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, καταλήγουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που χρησιμοποιούμε και νέε έννοιες, όπως για παράδειγμα ο εξυγχρονισμός της κοινωνικής ασφάλισης. Στο παρελθόν αυτό σήμαινε μάλλον τώρα σημαίνει τροποποίηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και σε μία γενικότερη πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση των συστημάτων αυτών, τα οποία αρχικά ήταν συστήματα καθαρά εθνικά και ήταν προφανώς συστήματα και προγράμματα αλληλεγγύης. Και κάτι ακόμα, εξίσου σημαντικό όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το Γιούρες, εταίρου στα πλαίσια του Γιούρες. Άκουσα την πρόταση την οποία κάνατε για μία επιτροπή ελέγχου, συντονισμού όλων αυτών των προγραμμάτων που συζητάμε. Εμεί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ω προς αυτό. Στα πλαίσια του Progress δεν υπήρξε ποτέ τέτοια επιτροπή. Υπήρχε μια ανεπίσημη μια άτυπη επιτροπή η οποία δεν λειτουργήσε για πάρα πολύ καιρό. Και εμείς είπαμε ότι τελικά δεν χρειαζόταν να υπάρχει και η επιτροπή αυτή. Κατά την άποψή μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ξεκάθαρη αρχή εταιρική σχέση, όπω και στα διορθωτικά ταμεία και όσον αφορά το Eures και απαντώ και στην κυρία Σρόντερ, δεν είναι αντίφαση να πούμε ότι θα προτιμούσαμε το Γιούρες και οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις Γιούρες να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε και αυτή τη βαθμιαία οπισθοδρόμηση υποβάθμιση του ρόλου μας στα πλαίσια του υφιστάμενου δικτύου και των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων. Και αν γίνει αυτό θα καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε την ισότιμη κινητικότητα των πολιτών. Ξέρετε ότι επί του παρόντος εξαιτία και των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών και εξαιτία κάποιων κακών νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων ιδίως όσον αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους και εξαιτία της μη συμμόρφωσης και της μη εφαρμογή της ε, ισότιμης μεταχείρισης στον χώρο εργασία, όπως αυτή προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, καταλήγουμε σε μια απορρίθμιση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και μια γενικότερη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν κανονικά την κοινοτικότητα των εργαζομένων. Το Eures είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδείξει ότι πραγματικά αξίζει, ότι πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε μια ισότιμη κινητικότητα των εργαζομένων και αυτό μπορεί να γίνει με την έντονη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστούμε πολύ, Κόνι Ρόιτερ. Ευχαριστώ. Προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση που είναι δύσκολη. Το δύσκολο είναι, το εύκολο είναι η στόχη όπως ανέφερε και η κυρία Σόντια. Ε, πράγματι, ποιος είναι κατά της μείωσης στόχιας. Αλλά βλέπουμε πως από τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα δεν έχουμε φτάσει τους στόχους των 20 εκατομμυρίων. Ποιο είναι κατά της ε, κοινωνικής ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικού διαλόγου. Βλέπουμε το, πως το κενό μεταξύ των πολύ πλουσίων και των πολύ φτωχών αυξάνεται. Δείτε την έκθεση που παρουσίασε η Κομισιόν ε, το Δεκέμβριο οι αριθμοί είναι εκεί πέρα και είναι σαφής. Οπότε το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, πρόγραμμα για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Κατόπιν, για την ε, κοινωνική καινοτομία. Το ερώτημα πάλι είναι το ίδιο. Ποιος είναι κατά της καινοτομίας. Τότε γιατί μιλάμε για κοινωνική καινοτομία. Γιατί μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία 15 χρόνια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητάμε αυτούς τους ωραίους γενικόλογους όρους. Απασχολησιμότητα, σας πενθυμίζω, ευελίξη ασφάλεια. Και πάντα δεν έχουμε ένα ορισμό τι εννοούμε, τι θέμε να πούμε εδώ πέρα. Και πρέπει να πω, μπορεί να είμαι αφελής, αλλά εξεπλάγει όταν έλαβα πρόσκληση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα συνέδριο για την κοινωνική καινοτομία και όταν διάβαζα το κείμενο πριν από δύο εβδομάδες αφορούσε ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ιαπωνικές πόλεις. Και είπα, μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Γιατί τι είναι η κοινωνική καινοτομία. Υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη, ανεργία, διακριτική μεταχείριση, α, μετανάστες ε, χωρίς ε, χαρτιά, ανεργία των νέων. Οπότε αυτό είναι να βρούμε απαντήσει για τις κοινωνικές μίκιο για να μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική και η καινοτόμος προοπτική είναι πως δεν θα επαναλάβουμε τα προγράμματα που λειτουργούσαν πριν από 20 χρόνια. Ούτε κανείς δεν είναι κατά της καινοτομία. αλλά βεβαίω θα βασιστούμε σε κοινωνικές ε, πολιτικές ε, οι οποίε βασίζονται σε στοιχεία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στο παρελθόν δεν κάναμε πολιτική με στοιχεία. Α, πάντων, δεν μπαίνω τώρα εγώ σε αυτή την πολεμική. Να περάσω τώρα σε κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει τη ε, συνεργασία. σω να μην ήμουν αρκετά συγκεκριμένο. Τι αφορά αυτό. Αφορά τη συνεργασία οπωσδήποτε των κοινωνικών εταίρων, αλλά και όσων δρούν στα προγράμματα κοινωνικής ε, συμπερίληψης και αφορά την ανάπτυξη, την εφαρμογή του προγράμματος, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Και ε, δώσαμε ένα παράδειγμα για το Progress. Ναι, πολλά από τα μέλη εποφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό. Ποιο ήταν το βασικό όφελος. Το να δικτυωθούμε και όχι βεβαίως να έχουμε μία εκπαίδευση με τη γαλλική έννοια της λέξης, αλλά μία ανάπτυξη των ικανοτήτων, γιατί πρέπει να διακρίνουμε το τι είναι η κοινωνία των πολιτών σε βορρά, νότο, ανατολή και δύση και νομίζω πως αυτό ε, σχετίζεται με την δυνατότητα αυτών των οργανώσεων να βρουν απαντήσεις να είναι καινοτόμες ή λιγότερο. Οπωσδήποτε όμως αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του Progress. Επίσης ρωτήσατε κυρία Στάινροκ το τι άποψη έχουμε για το ότι έφυγε η η αντιμετώπιση των διακρίσεων. Ε, δεν, το, δεν μας άρεσε κιόλα. γιατί ε, αυτά πάνε μαζί με την κοινωνική συμπερίληψη. Εσείς ψηφίζετε εδώ πέρα τη σύσταση περί συμπερίληψης και βέβαια αφορούσε τρία στοιχεία ενεργητικές πολιτικές εργασίες αγοράς, ελάχιστο εισόδημα, κοινωνικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα είχε και το ζήτημα των μη διακρίσεων γιατί απέχουμε ακόμα από την αρχή ίσης πληρωμής ε, για ίδια εργασία. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα για να μην ε, χάσουμε την προσθέμενη αξία του Progress και για να έχουμε την δυνατότητα πραγματικής ε, απάντησης στις κοινωνικές ανάγκες για την επιχειρηματικότητα. Εάν την επιχειρηματικότητα την εννοούμε με τη γαλλική έννοια του να επιχειρεί κανείς κάτι, κανείς δεν είναι κατά. Αυτό κάνουν οι κοινωνικές ΜΚΟ. Αλλά εάν είναι μόνο από την πλευρά των επιχειρήσεων και να λέμε μόνο οι επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε είναι πρόβλημα γιατί όπως ξέρετε παλεύουμε και για την αναγνώριση του ζητήματος ε, των ε, κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Οπότε είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Συγκεκριμένα ερωτήματα της Ελίζα Στρέτερ για το αποθεματικό. Πράγματι σε 7 χρόνια ε, λέμε πως ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια θετική ευελιξία για να βρεθούν κάποιες απαντήσεις στον τομέα αυτών, αλλά το ζήτημα είναι ποιος το διοικεί, το κάνει μόνο η Κομισιόν ή είναι πραγματικά ένα συντονισμός του προγράμματος που βασίζεται σε πραγματικές ε, σχέσεις ε, συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών τότε να, το μιλήσουμε, να μιλήσουμε γι' αυτό. Και νομίζω πως υπάρχει πράγματι η δυνατότητα για καινοτομία, αλλαγή και συγκεκριμένες λύσεις, γιατί ναι, το πρόγραμμα αυτό έχει στόχους με τους οποίους συμφωνούμε, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, αν και έχουμε τη γενικότερη εντύπωση ότι μόλις την ξεκινάμε. Προφανώς θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Μας κατατόπισαν σίγουρα οι ομιλητές μας. Ξέρουμε πλέον ποιος είναι ο ρόλος μας, ο ρόλος αυτής της Επιτροπής και με τη βοήθεια της εισηγήτριάς μας θα προσπαθήσουμε να τοποθετηθούμε σχετικά με τη θέσπιση αυτού του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελικά θέτει και αρκετά προβλήματα και πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε και με την ουσία του προγράμματος αλλά και τη διάρθρωσή του σε αυτούς τους τρεις άξονες. Πώς θα καταφέρουμε να τους συμπεριλάβουμε σε ένα ενιαίο κείμενο. Αν επιθυμεί κάποιος άλλος να πάρει το λόγο εισηγήτρια, σύντομα παρακαλώ. Und den äh, Fragestellerinnen und Fragestellern heute danken, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους έθεσαν ερωτήσεις γιατί είχαμε ε, σημαντικές προτάσεις, ποια είναι τα ανοιχτά σημεία που πρέπει να γίνουμε πιο ξεκάθαροι στους ορισμούς έτσι ώστε ε, όλοι να ε, διευκολυνθούμε στην εργασία μας. Η αρχή της συνεργασία με ναι, τους κοινωνικούς εταίρους στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα είναι ο διαχωρισμός και ακριβώς αυτό το δείχνει το ζήτημα όηρες. Δείχνει πόσο ε, σημαντικές ε, είναι οι επιπτώσεις αν κάνουμε ε, λάθη και πράγματι είχα σκεφτεί και εγώ πως ε, καλύτερα ήταν το ΟΙΡΕΣ να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αλλά μετά διαπιστώνουμε πως ε, χάνονται σημαντικά κομμάτια του ΟΙΡΕΣ, π.χ. συνοριακές συνεργασίες, γιατί είναι σε διαφορετικά κρατημέλη που έχουν άλλες προτεραιότητες. Όταν μιλάμε για διασυνοριακές συνεργασίες, πρέπει να έχουμε ενιαίους στόχους. Εάν δεν τους έχουμε αυτούς, δεν υπάρχουν. Οι διασυνοριακές συνεργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές στην κινητικότητα των εργαζομένων. Το μεγαλύτερο κομμάτι των Ευρωπαίων εργαζομένων που δεν δουλεύει στη χώρα του δουλεύει σε διασυνοριακές συνεργασίες. Νομίζω λοιπόν πως θα ήταν μεγάλο λάθος να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι από εδώ πέρα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ακριβώς για τους ε, εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, τις εργασίες μας και το επόμενο στάδιο είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης της κυρίας ε, Στάνμπρουκ το Μάρτιο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστούμε θερμά τους καλεσμένους μας και θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τους ομιλητές μας στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης όπου θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με αρκετούς ε, παρεμβαίνοντες όσον αφορά τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρωτού δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, η οποία θα κάνει μια πρώτη εισαγωγή και θα κατευθύνει λίγο τις ερωτήσεις που θα κάνουμε στους ομιλητές μας. Να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ σήμερα το απόγευμα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση ως προς το ΕΚΤ και όλοι ενδιαφέρονται από τους πανελίστ που έχουμε εδώ. En fait, euh, dois dire que euh, Η εξέλιξη του ΕΚΤ έχει μεγάλη σημασία και βλέπουμε ότι η προηγούμενη συζήτηση έχει σημεία διασύνδεσης με προγράμματα που αφορούν στόχους του ΕΚΤ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική και επαγγελματική συμμετοχή είναι ύψιστη της σημασία σήμερα. Ένα από τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσει είναι η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ και η εφαρμογή προγραμμάτων in situ. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή θέληση κοινωνικής συμμετοχής και ενσωμάτωσης. Τι σύνδεση λοιπόν υπάρχει με τις πολιτικές που τίθενται σε εφαρμογή τοπικά για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ένα δεύτερο θέμα εξίσου σημαντικό βλέπουμε ότι η ρήτρα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας έχει μεγάλη σημασία για την ε, εδαφική εφαρμογή. Nous sommes extrêmement intéressés à travers le témoignage des Και γι' αυτό θα μας πούνε και οι εμπειρογνώμονες ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι πώς να αυξήσουμε τις επαγγελματικές αρμοδιότητες του συνόλου των μισθωτών και εκτός και εντός εργασίας και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν ισχυρά επαγγελματικά προσόντα, για να μην αποκλειστούν κυρίως οι νέοι από την κοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν με έναν ευρύ ορίζοντα και οι εμπειρογνώμονές μας θα μας κατευθύνουν έτσι ώστε να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ανδρέας Μπάρτελ, υπεύθυνο επί ευρωπαϊκών θεμάτων από το Arbeiter Wohlfahrt Bundesverband. Verband. Ε, σας δίνω λοιπόν το λόγο να μας αναπτύξετε το θέμα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να σας πω κάποια πράγματα σήμερα. Μου ζήτησαν να πω κάποια πράγματα για το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και το πού θέλουμε να πάμε. Προσπαθήσατε να πείτε από πού ε, προέρχομαι. Είμαι λοιπόν από την Ένωση ε, πρόνοιας εργαζομένων, ε, μια δευτεροβάθμια οργάνωση. Ε, υπάρχει και η Κάριτας, βεβαίως μεγαλύτερη από μας. Καλύπτουμε με 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας στη Γερμανία. Εγώ ο ίδιος εδώ και 16 χρόνια δραστηριοποιούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 10 χρόνια ε, εργαζόμουν στα έργα και 6 χρόνια στον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι τώρα. Πώς έχει η κατάσταση στη Γερμανία. Ξέρετε πως πέρα από ένα ομοσπονδιακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουμε και 16 ε, προγράμματα στα κρατήδια και διάφορα άλλα. Υπάρχουν λοιπόν κάτω από αυτά 61 υποπρογράμματα με τα οποία εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς και οι, διάφοροι αυτοί, οι διάφορες προενιακές ενώσεις έχουν ε, ένα πρόγραμμα με το ωραίο όνομα Ούριος Άνεμος το οποίο βασίζεται σε ένα άρθρο του τωρινού κανονισμού. Τι κάνουμε λοιπόν. Κυρίως ασχολούμαστε με τα μέτρα για την εξέλιξη του προσωπικού, για την προληπτική υγεία, για την διαβίου εκπαίδευση και βεβαίως ένα γενικό θέμα του πώς μπορούμε να έχουμε ένα προγραμματισμό σταδιοδρομίας και τα λοιπά. Οι βασικοί χρήστες είναι οι εργαζόμενοι του τομέα της βοήθειας των ηλικιωμένων, των παιδιών και των αναπήρων. Όλος αυτός ο τομέας, δηλαδή της κοινωνικής πρόνοιας. Στη Γερμανία συμβαίνει το εξή, η κοινωνική οικονομία είναι ένας κλάδος με ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να πω πως η δημογραφική αλλαγή καλύπτει όλες τις χώρες και υποθέτουμε πως μέχρι το 2030 θα έχουμε ε, θα χρειαζόμαστε 75% περισσότερους εργαζομένους, το οποίο από πού θα προκύψουν το μεγάλο ερώτημα, γιατί βεβαίως μεγαλώνουμε, αλλά έχουμε λιγότερες δυνατότητες για προσλήψεις και βεβαίως πρέπει να διατηρήσουμε και τα άτομα τα οποία έχουμε ήδη στον τομέα αυτών. Όπως είπα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γερμανίας Εργασίες με και Κοινωνική Ασφάλισης της Γερμανίας εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ανέφερα. Πώς έγινε αυτό. Έχουμε ε, ζητήσει και λάβαμε τεχνική αροχή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είχαμε επίσης ένα ε, μια υπηρεσία στήριξης για την εφαρμογή του προγράμματος και μια ομάδα καθοδήγησης όπου συμμετέχει ισότιμα και ο δημόσιος τομέας και οι ενώσεις μας και έτσι καθοδηγείται επί της ουσίας το πρόγραμμα και τα διάφορα έργα. Και, όπως σας είπα, η υπηρεσία αυτή είναι αρμοδιακή και για την παρακολούθηση, κάτι περισσότερο δηλαδή από την αξιολόγηση, θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ε, πτυχές ε, ε, διαρκής ή όχι. Ο όγκος του προγράμματος ήταν μικρός, γύρω στα 60 εκατομμύρια μετά από έξι προσκλήσεις ε, εξαντλήσαμε το ποσό, αλλά βεβαίως τα έργα θα συνεχιστούν μέχρι το 2014. 134 έργα εντάχθηκαν. Οπότε, τι ε, προβλέπουμε για, τον για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο για να δούμε και το τι εννοούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για εμάς είναι ένα εργαστήριο όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε νέες ιδέες. Αυτό για εμάς ήταν άξιση της απασχολησιμότητας αλλά και το ζήτημα βεβαίως της μείωσης της στόχιας ήταν κάτι το σημαντικό να μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες. Δεν θέλουμε να εκπληρώσουμε βασικές αρμοδιότητες των, των, αυτών τα θα έπρεπε να κάνει το κράτος ούτως ή άλλως, απλά αν υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να προετοιμαστούν ή να κρατήσουν τη δουλειά τους, να τους βοηθήσουμε. Από εκεί προκύπτουν και οι ιδέες που έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική του 2020 και είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς, αλλά βεβαίως κοιτάμε και πάρα πολύ και το εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στη Γερμανία, σε ποιο βαθμό ε, επιτυγχάνει αυτούς τους ε, στόχους. Χτες ε, λοιπόν λάβαμε την ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το πώς δηλαδή μπορούμε να εφαρμόσουμε το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και δυστυχώς δεν περιέχει τα πράγματα τα οποία θα θέλαμε, ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση τη στόχια, αλλά εξακολουθούν να κολλάνε σε ένα δίκτυ στη Γερμανία και παραμελούν τα υπόλοιπα. Ανεξαρτήτω από αυτό βεβαίως ε, κοιτάμε το ποιοι θα είναι οι κλάδοι που θα έχουμε ανάπτυξη στο μέλλον για να μπορέσουμε να δούμε τη δημογραφική αλλαγή, μεγάλο κομμάτι θα είναι βεβαίως η φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν είναι το κατ' αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι νομίζω γνωστό, αλλά και αυτός είναι ο άλλος σημαντικός στόχος πολέμηση της φτώχειας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι κάτι τόσο σωστό και θετικό και έτσι θα πρέπει να παραμείνει και δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί δηλαδή προσπάθειες του Συμβουλίου για να διαγραφεί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απορρίψουμε. Τώρα όσον αφορά τη μακροοικονομική διάσταση αναφέρθηκαν ήδη κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς είναι απλά να υπάρξει περικοπή ε, όταν δεν πάνε καλά τα μακροοικονομικά πράγματα. Ειδικά ε, χωρίς να γίνει μια αξιολόγηση του αντικτύπου. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν προγράμματα για τους άστεγους, ε, φυλακισμένους ε, κλπ. να κόβονται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στα οικονομικά. Πρέπει να γίνει μια μελέτη κοινωνικού αντικτύπου για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με αυτές τις ομάδες στόχους. Είχαμε λοιπόν ε, επεξεργαστεί κάποιους κοινωνικούς δείκτες για το θέμα αυτό ακριβώς, γιατί θεωρούμε πως δεν επαρκεί να έχουμε μόνο οικονομικούς παράγοντες ε, για την κατανομή των κονδυλίων του ΕΚΤ, ειδικά όσον αφορά το θέμα φτώχεια. Η αρχή αυτή της συνεργασίας επίσης αναφέρθηκε, είναι κάτι το οποίο εμείς το στηρίζουμε πάρα πολύ, δεν το χρειαζόμαστε βεβαίω μόνο για τους κοινωνικούς εταίρους. Χαιρόμαστε για το ότι στην διατύπωση αναφέρονται η ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών. Αυτό για εμάς είναι ουσιώδες γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και αυτό το οποίο είπα είναι πως η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι συνομιλία σε ίσο επίπεδο και να μην λαμβάνουμε ε, διαταγές και εκ των υστέρων έγκριση των αποτελεσμάτων. Παραδείγματο χάρη οι επιτροπές παρακολούθησης στη Γερμανία ε, εγκρίνουν εκ των υστέρων τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο των προγραμμάτων. Γι' αυτό εξετάζουμε πότε θα έρθει ο κώδικας συμπεριφοράς της ε, Κομισιόν ε, που θα διαμορφώσει ε, ουσιαστικά και ποιοτικά τα προγράμματα αυτά. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες ιδέες και ελπίζουμε ακριβώς να υπάρξει αλλαγή στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Οπότε τώρα, στην πράξη, το τι γίνεται μπορεί να υπάρξει μια απλοποίηση όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, το θέμα των καταποκοπήν ποσών, ε, μεγαλύτερη επίσης ευελιξία στο ποσοστό συγχρηματοδότηση στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και επίσης το ζήτημα της τεχνικής ε, αρρωγής είναι επίσης σημαντικό αν είναι να οικοδομήσουμε την διοικητική ικανότητα θα πρέπει βεβαίω να υπάρχει η ικανότητα να απορροφηθούν αυτά τα λεφτά και αυτό άρα σημαίνει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε όχι μόνο τις περιοχές που δεν είναι ανεπτυγμένες, αλλά και οι περιοχές οι οποίες είναι σε μια μεταβατική φάση για να χρηματοδοτηθούν. Και ο, επειδή ο χρόνος πιέζει σύντομα το τι σκεφτόμαστε για το μέλλον, έχουμε δύο μεγάλους θεματικούς τομείς. Ο ένας είναι ε, διαμόρφωση της δημογραφικής αλλαγής μέσω ενίσχυσης κοινωνικής οικονομίας. Δεύτερον, καταπολέμηση της φτώχειας. Εκεί πέρα θεωρούμε πως πρέπει να γίνει κάτι επιγόντως στη Γερμανία θα αναφερθώ λίγο στις ε, προτεραιότητες ε, των ε, επενδύσεων να υπάρξει δηλαδή καταπολέμηση της στόχιας κοινωνική ενσωμάτωση. Είμαστε σε συνομιλία με την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε η συνεργασία να ακολουθείται όπως θα έπρεπε από πλευράς ομοσπονδιακού κράτους. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα μηνύματα για τον κανονισμό αυτό, έτσι ώστε και μια χώρα όπως η Γερμανία να μην μπορέσει να αποφύγει αυτή την συνεργασία που επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Εργετιάν, Γενικό Γραμματέα Περιφερειακών Υποθέσεων στην ομαρχία Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω την καθημερινή πραγματικότητα της διαχείρισης των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή η οποία είναι κυρίως αγροτική μέσων διαστάσεων, η περίφημη περιοχή Πατού Σαγόντα στη Γαλλία. Ένα μέρος της διαχείριση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γίνεται από τον ιατρικό κράτος και ένα άλλο μέρος των κονδυλίων τυχαίνει διαχείρισης από την περιφέρεια Πατού Σαγόντα, σε τοπικό περιφερειακό δηλαδή επίπεδο. Η αγροτική λοιπόν αυτή περιοχή έχει 125-127 εκατομμύρια ευρώ για 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή ένα 2,7% του συνολικού πληθυσμού της Γαλλίας. Κατά 89% βρισκόμαστε κοντά στον μέσο, στο μέσο κοινοτικό ΕΠΑ και οι βασικότερες δραστηριότητες είναι αγροτικές. Εξάγουμε προϊόντα όπως το κονιάκ και διάφορα μεταποιημένα προϊόντα, τα οποία προέρχονται από τον αγροδιατροφικό τομέα. Η περιφέρεια αυτή, όπως και άλλες μεγάλες περιφέρειες της Γαλλίας, επλήγει από το 2008 και μετά από την γενικότερη οικονομική κρίση και πιο συγκεκριμένα από το καλοκαίρι του 2011 και μετά. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοηθά ιδιαίτερα τις γαλλικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι υπάρχει μια σύμβαση εμπιστοσύνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για να εφαρμοστούν δηλαδή συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές επίσης στον τομέα του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης. 9,3% είναι η ανεργία στην Γαλλία, 8,9% στην περιοχή Πατού Σαγόντα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Θέλουμε προφανώς να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρύνουμε την επιστροφή στη θέση, σε θέσεις εργασίας των ανθρώπων αυτών οι οποίοι είναι άνεργοι. Στον χρόνο που έχω θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε μια μικρή περιφέρεια αλλά υποφελούμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πλήρως. Κατά ένα 72% χρησιμοποιούμε τους πόρους του ταμείου αυτού. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 90 εκατομμύρια δίνονται συγκεκριμένα στην δική μας την περιοχή για την πραγματοποίηση πάρα πολλών προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά έχουν ένα προπολογισμό γύρω στα 51 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερη σημασία που δίνει η περιοχή Πουατού Σαγόντ στα κοινωνικά έργα, στα κοινωνικά προγράμματα τα οποία προωθούνται και τα οποία θα σας περιγράψω και στη συνέχεια της παρουσίασής μου. Όπως σας είπα, η πολιτική απασχόληση στη Γαλλία αποφασίστηκε σε κεντρικό επίπεδο, αλλά η διαχείριση κατά 80% γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Αναφέρομαι στο 80% των κονδυλίων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εδώ και κάποια χρόνια το κράτος έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης των πιο φτωχών πολιτών, δίνοντάς τους τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να ξαναβρούν μια θέση εργασίας και προκειμένου να σε θέση να ζήσουν αξιοπρεπώς και να καταφέρουν να χρηματοδοτήσουν τη δραστηριότητά τους είναι οι διαφορετικοί νομοί στην, η στη Γαλλία που χειρίζεται το πρόγραμμα αυτό και εμεί στη δική μας την περιφέρεια βοηθούμε τους τέσσερις νομούς που υπάγονται στην Πουατού Σαγόντα δίνοντας 3 με 4 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε διάφορα προγράμματα ε, κοινωνικής ένταξης όπου βοηθούμε πολλούς πολίτες να επιστρέψουν στην εργασία, να ξαναβρούν μια δουλειά. έχουμε και ένα παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όπου 10.500 άτομα που φελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό και ένα 60% των ατόμων κατάφεραν να ξαναβρούν δουλειά. Δημιουργία θέσεων εργασίας, επιστροφή στην εργασία, καταπολέμηση επίσης της πρόορης αποχώρησης από το σχολείο. Προσπαθούμε λοιπόν τα προγράμματα αυτά να βοηθήσουμε τους πολίτες σε όλες τις ηλικίες να αποφεληθούν από τα προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο λοιπόν χρηματοδοτεί κάποια συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι διυπουργικά τις περισσότερες φορές και μέσω της χρηματοδότησης αυτής προσπαθούμε να βοηθήσουμε για την καταπολέμηση της πρόορης αποχώρησης από το σχολείο, δίνουμε συγκεκριμένες, ε, προωθούμε συγκεκριμένα προγράμματα για την ε, κατάρτιση των νέων. Έχουμε διάφορα τέτοια κέντρα σε διάφορα μέρη της περιοχής που Σαγόντε. Και έχουμε ένα 80% των νέων τελικά που έχουν εγκαταλείψει με το σχολείο, αλλά καταφέρνουν να παρακολουθήσουν διάφορα προγράμματα κατάρτισης και τελικά να βρουν μια θέση εργασίας. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε επίση τον αναλφαβητισμό, ζήτημα για το οποίο μιλάμε πάρα πολύ. Περίπου 5 εκατομμύρια είναι αναλφάβητοι στη Γαλλία. Στην Πρατούσα Αγών προφανώς υπάρχουν αναλφάβητοι και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτούς να ανακτήσουν κάποιες βασικές γενικές γνώσεις και Έχουμε πάλι εδώ πέρα κάποια ειδικά προγράμματα προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτούς να καταφέρουν να ανακτήσουν κάποιες δεξιότητες για να βρουν στη συνέχεια μία θέση εργασίας. Προσπαθούμε στην περιοχή Πατιού Σαγών να αντιμετωπίσουμε από τη μια τις οικονομικές αλλαγές, να προσαρμοστούμε στις οικονομικές αλλαγές. Στη συνέχεια προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανέργους, όπως σας είπα, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την κοινωνική ένταξη. Όσον αφορά τώρα τις οικονομικές αλλαγές και την υποστήριξη, τη δημόσια υποστήριξη για τους πολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ένα 80% του επιχειρησιακού προγράμματος της Πατού Σαγόντα δίνεται για το πρόγραμμα αυτό και ένα περίπου 50% δίνεται για το άλλο πρόγραμμα το οποίο σας περιέγραψα. Προσπαθούμε να αποστοκοπήσουμε και να αποτιμήσουμε τα προγράμματα αυτά με τη βοήθεια του κεντρικού κράτους αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε ένα σύστημα πληροφόρησης το οποίο έχει αρχίσει να ισχύει εδώ και κάποια χρόνια, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε μία ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτό γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά μπορούμε να έχουμε και μία κάποια, ένα κάποιο διάλογο διαχείρισης, διακυβέρνησης ανάμεσα στο, στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε σε εθνικό επίπεδο συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και κάτι άλλο. Συγχρηματοδοτή και με άλλες περιφέρειες όπως η Ρον Αλπ και η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Υπάρχει λοιπόν ένας οικονομικός άξονας μέσω ΕΚΤ και Υπάρχουν διάφορα επίπεδα προγραμματισμού, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχει προγραμματισμός, διότι μιλάμε για ένα 53% ε, προγραμματισμού αυτού του επίπεδου και γι' αυτό στα πλαίσια αυτής της ένταξης μπορούν να βρουν ε, θέσεις εργασίας στο 1 τρίτον των ετούντων. Κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Εντάχει θα ήθελα να σας πω, να μιλήσω για ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές ε, οι οποίες προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τις προτεραιότητες γύρω από τρεις ε, άξονες. Να προετοιμάσουμε τους ε, εργαζομένους ε, γύρω από τους οικονομικούς άξονες. Επίσης, να προετοιμάσουμε τους νέους για εργασία μακριά από τον τόπο διαμονής και γενικότερη προετοιμασία για ανταπόκριση σε νέες θέσεις εργασίας όπου και αν βρίσκονται αυτές. Θα πρέπει λοιπόν και ο ενεργός και ο μη ενεργός ε, πληθυσμός να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο το οποίο οργανώνεται επιτοπίως για να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ε, εδαφική ανάπτυξη της εργασίας. Όπως γίνεται στη Γαλλία, στη Γαλλία επίσης υπάρχουν και οργανισμοί διαμεσολαβητές για τη έβρεση εργασίας. Πιστεύω ότι σήμερα θα πρέπει να απλουστεύσουμε τον επίσημο έλεγχο του επιχειρησιακού σχεδίου και αυτό μέσα στα πλαίσια και του ΕΚΤ. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την χρήση των ταμείων και για σχέδια και για ε, πιο μικρούς οργανισμούς, όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Γερμανία. Γιατί να μην υπάρχει ένα εγχειρίδιο διαχείρισης και για τους χρήστες του ΕΚΤ, έτσι ώστε να μετρήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα και τους στόχους. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη χρήση και καλύτεροι δείκτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα και να είχαμε και ένα διευρυμένο ΕΚΤ όπως ισχύει για την ε, διατροφική βοήθεια, για τους πλέον φτωχούς, θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το ΕΚΤ και να έχουμε καλύτερες ε, διαρθρώσεις και αυτό αφορά και το ε, Ταμείο Προσαρμογής την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να βρούμε πασαρέλες για μελλοντικές επιχειρησιακές δράσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τιέν. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Άνταμ Κούλμαν, ο οποίος είναι υπεύθυνο πολιτικής του Open Society Institute από τη Βουδαπέστη έχετε το λόγο. Έχετε γύρω στα 10 λεπτά. Ε, ο χρόνος πιέζει. Αλλά όπως είπα, θέλω να απευθύνω έκκληση και στους τρεις σας, αν έχετε κάτι γραπτός. Και εγώ η ίδια είμαι σκιοδησυγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οπότε, σας παρακαλώ, δώστε τα στην γραμματεία ή δυνατόν και σήμερα για να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις σας. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Κούλμαν λοιπόν. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα για το πρόγραμμά μας. Δεν χρησιμοποιούμε μόνο το ΕΚΤ, συν ε, χρηματοδοτούμε και εμείς για να έχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις για ΜΚΟ. Ε, εργαζόμαστε στη δημοκρατία της Τσεχίας, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σλοβακία εκτός από την ε, Ουγγαρία. Θα ομαδοποιήσω τα μηνύματά μου σε τρεις κατηγορίες. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή έκανε μια πολύ καλή πρόταση που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα. Πιστεύουμε ότι μερικά από αυτά θα υποστηριχθούν και από το Συμβούλιο και άλλα ίσως όχι και τόσο πολύ. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλειών και του Κοινοβουλίου. Uh, uh, Όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη χρήση των ταμείων και πιστεύουμε ότι τα ταμεία είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή στοχοθέτηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσει και το Συμβούλιο. Έχει μεγάλη σημασία για να δούμε πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ένα χρόνο πριν για την χαρτογράφηση των περιοχών φτώχειας, τους υπόψη και τους Ρωμά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσω ότι η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ θα έχει μεγαλύτερη σημασία περισσότερο από το ΕΚΠΑ, γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα επιμέρους ζητήματα. Ποια είναι τα ζητήματα λοιπόν αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά στα πλαίσια του σχεδίου πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήματα τα οποία δεν υποστηρίζει επαρκώς πιστεύω ο άλλος συνομοθέτης, δηλαδή το Συμβούλιο. Πολλοί ήδη αναφέρθηκαν στα κονδύλια αυτά τα οποία θα πρέπει να δοθούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για ζητήματα όπως ε, η κοινωνική ενσωμάτωση, η κοινωνική ένταξη. Επίσης, όσον αφορά την αιρεσιμότητα, πολλά πράγματα έχουν ήδη υποθεί για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στην ε, κοινωνική αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη τελικά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εξάντε αιρεσιμότητα, που σημαίνει δηλαδή ότι ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν κάποια προκατακτικά προγράμματα για την ε, χρησιμοποίηση των πόρων. Αυτό θα είναι πολύ θετικό για τη σωστή χρησιμοποίηση των πόρων αυτών. Όσον αφορά την ε, κοινωνική ενσωμάτωση, την ενσωμάτωση των Ρωμά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές προϋποθέσεις, οι οποίες να ισχύουν για την κατανάλωση, για τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων, των κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης πιστεύω ότι το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να έχει κάποιες θεσμικές εγγύησεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης των υπαλλήλων εκείνων που εργάζονται στον τομέα της κατανομής των κοινωτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να λέγεται στον κανονισμό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για την πρόθεση των ίσων ευκαιριών και ότι θα υπάρχουν κάποιες σχετικές ε, δραστηριότητες. Και συμφωνώ με όσους ε, ήδη είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε μια οικοδόμηση ικανοτήτων για τους εταίρους και έναν κώδικα συμπεριφοράς. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που πιστεύω ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Καταρχάς, όσον αφορά την εξάντε αιρεσιμότητα. Η διατύπωση του κανονισμού λέει ότι θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένε στρατηγικές. Δεν είναι σαφές όμως αν οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει ήδη να έχουν αρχίσει να ισχύουν αν θα πλαισιώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω θα πρέπει να λέγεται ρητός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει συγκεκριμένη εντολή. Επίσης, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ρωμά επί του παρόντος αποτελεί μέρος της εξάντερες ημότητας για την κοινωνική ένταξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κάποια προγράμματα ενσωμάτωση στον Ρωμά, όπου λέγεται συγκεκριμένα ότι η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων στέγασης, απασχόλησης, ε, υγειονομικής περίθαλψης κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, το συγκεκριμένο ζήτημα των Ρωμά να ενταχθεί στις, ε, στην κοινωνική αιρεσιμότητα και θα πρέπει συγκεκριμένα να προβλέπονται τα προγράμματα αυτά για την εκπαίδευση, την στέγαση και το Πέρυσι το Μάρτιο είχαμε ήδη πει ότι τα διεθνωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξάλληψη της, του κοινωνικού διαχωρισμού και για την πρόθεση των ίσων ευκαιριών. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να θέσει ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω μάλιστα στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τονίσει τις προϋποθέσεις αυτές, αλλά τελικά δεν ενσωματώθηκαν στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης οι θεσμικές εγγυήσει θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει στην δομή της χρήσης των ταμείων αυτών και της διαχείρισης των ταμείων ένα άτομο το οποίο είναι πραγματικά υπεύθυνο για την, για την εφαρμογή, την τήρηση αυτών των κοινωνικών προϋποθέσεων. Αυτά είχα να σας πω και έχω ήδη στείλει γραπτό στις συγκεκριμένες μου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, ε, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Γκέντς έχει το λόγο. Χαίρομαι που άκουσα τα σχόλια γιατί συμβαδίζουν με τη δική μας λογιστική. Εδώ στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Συμφώνω με τον κύριο Μπάρτας, ο οποίος είπε ότι ένας ε, βασικός στόχος είναι να αντισταθούμε στο Συμβούλιο. Κάτι το οποίο τόνισε και ο κύριος Κούλμαν. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη την ε, κοινωνική συμμετοχή και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το περιφράξουμε κάπως γιατί διαφορετικά ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Συμφωνούμε με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, κάτι το οποίο μιλά για ε, μεταχείριση αυτών, ειδική μεταχείριση αυτών που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ε, ναι, μιλάμε για μείωση, καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Εγώ θα είμαι εισηγήτρια στο ΛΥΜΠΕ για αυτά τα προγράμματα ηθαγένειας που αφορούν και την εξάλληψη των διακρίσεων. Άρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε αυτούς τους κανονισμούς σε σχέση με το γενικό κανονισμό, ο οποίος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ορισμένα κράτη τα οποία την χάνουν υποστήριξης από αυτά τα προγράμματα και την Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και ποιος είναι ο στόχος ως προς την αρχή της ε, εταιρικότητας δεν πρέπει να το δούμε μόνο από πλευρά σκεπτικού, θα πρέπει να το δούμε επιχειρησιακά. Να βρούμε κατευθυντήριες γραμμές, γιατί θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις ο κύριος Κούλμαν μίλησε για αυτές τις διακρίσεις, γιατί το πραγματικό θέμα είναι η εφαρμογή όλων αυτών των κανονισμών. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε την έλλειψη πολιτικής θέλησης, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, για να έχουμε εγγυήσεις για την εφαρμογή ε, παρόμοιων έννοιων. Βλέπω ότι αναφέρθηκαν πολλά και χρήσιμα. Και όπως είπε και η Ελίζαμπεθ, θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτα και όλα τα γραπτά σχόλια κατά τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να δώσω λόγο στην εισηγήτρια και δεν ξέρω νομίζω ότι έχετε και μία ερώτηση, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές μας. Οι παρεμβάσεις τους αλληλοσυμπληρώνονται και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν θα αναφερθώ σε ερωτήσεις που έθεσε η Κίνγκα Μπόνς, αλλά πάντως θα συνεχίσω μετά τις ερωτήσεις αυτές. Προκειμένου να επιδείξουμε μία επικοδομητική στάση, είναι σημαντικό να συντοπίσουμε ότι μιλάμε όλο και περισσότερο για την βούληση που υπάρχει να αναλάβουμε δράση επιτόπου. Μπορείτε όμως να μας δώσετε κάποιες συμβουλές όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες πάνω στους οποίους θα μπορούσαμε να στηριχτούμε προκειμένου να αποτιμήσουμε την αποδοτικότητα ορισμένων πολιτικών όχι μόνο για να μετρήσουμε την αποδοτικότητά τους αλλά για να κινητοποιήσουμε και τους αρμόδιους φορείς να γίνουν λίγο πιο αποτελεσματικοί επιτόπου έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά ταμεία να δημιουργήσουν μια θετική επίπτωση μόχλευσης. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερον, Εκτίμησε ιδιαίτερα ότι πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε περιόδους μεταβατικές. Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά που εφαρμόσουμε κοινοτικές πολιτικές να έχουμε τις μεταβατικές αυτές περιφέρειες και μας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, περιοχές που ουσιαστικά εποφελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν υπάρχουν όμως πάρα πολλά προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πολλές φορές σε επίπεδο περιφέρειας υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα, πολλά διαφορετικά προγράμματα τα οποία δεν απαιτούν όλα σημαντική, πολύ ψηλή χρηματοδότηση. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να πλουστεύσουμε την υφιστάμενη αυτή κατάσταση, το ότι πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα προγράμματα αυτά, τα οποία επιτόπου κανείς πρέπει να εφαρμόσει. Τρίτον, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, είπατε ότι το κοινωνικό ταμείο μπορεί να υποστηρίξει κάποια καινοτόμα προγράμματα προγράμματα κατάρτισης τα οποία συμπληρώνουν κάποιες εθνικές πολιτικές. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί τελικά να βοηθήσει περισσότερο τις κρατικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος. Νομίζω θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την τάση αυτή. Τέταρτον, πολλοί αναφέρθηκαν στο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προβλέψουμε κάποια προγράμματα και ότι, για παράδειγμα, στην απασχόληση όσον αφορά τις θέσεις εργασίας δεν, δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με, τη με την δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και με τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσατε πάλι να μας δώσετε κάποιες πρώτες ιδέες έτσι ώστε στις επόμενες φάσεις των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να καταφέρουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί το ζήτημα αυτό. Αυτές είναι ερωτήσει μου, κυρία Πρόεδρε. Ähm, Πρόεδρος, και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα ερωτήματα, γιατί και εγώ είμαι σκιώδης. Ähm, και με έχει απασχολήσει αυτός ο κανονισμός σε επίπεδο λεπτομέρειε. Πρώτον προς τον κύριο Μπάρτελς. Υπάρχει το άρθρο 6 ε, που τάσεται υπέρ α, της αρχής της εταιρικότητας. Όμως εδώ υπάρχουν ε, πολλά στρώματα εταιρικής υποστήριξης. Θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε περί αυτού, γιατί εγώ αντιτάσσομαι. Θεωρώ ότι οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη ανεξάρτητα από τα κράτη που αφορούν. Και η αρχή της εταιρικότητας δεν είναι τόσο καλή στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να πούμε ότι δεν θα πρέπει να τύχει υποστήριξης. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση. Προς τον κύριο Ετιέν. Ansatz haben des des ESF würde mich interessieren, wie Sie diese Έχετε ε, μιλήσει, μιλήσατε μάλλον για το ΕΚΤ και τον τοπικό ρόλο, το ρόλο των, της τοπικής, των τοπικών αρχών. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με τον κανονισμό του ΕΚΤ. Εμείς μιλάμε για μία ρήτρα 5% από πλευράς της ομάδας των Πρασίνων. Το είδαμε και για την αστική συνεργασία, στο Λίντερ, στην περιφερειακή ανάπτυξη και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της απασχόλησης. Υπάρχει κάποιος άλλος, όχι δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές έχετε το λόγο πέντε, για πέντε λεπτά ο καθένας, γιατί θέλουμε να δώσουμε το λόγο και στην Επιτροπή στη συνέχεια. Σας ακούμε έναν έναν. Με την αντίστροφη σειρά ο κύριος Κούλμαν. Ετιέν και Μπάρτελς. Κύριε Κούλμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ως προς την ε, μέτρηση της προόδου, ε, δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόμαστε εθνικούς δείκτες. Πρωτίστως υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να μετρήσουμε τις βελτιώσεις και τη βελτίωση γενικότερα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε δείκτες. Δηλαδή αν έχουμε το χάρτη κρίσης ή τη χαρτογράφηση φτώχειας βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε αυτές τις περιφέρειες. Θα πρέπει όμως να έχουμε και συλλογή ενδεχομένως εθνικών δικτών. Ως προς την απλούστευση, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο κανονισμός να είναι σαφής. Ο τρέχον κανονισμός ενέχει δυνατότητες απλούστευσης αλλά υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας και γι' αυτό πιστεύω ότι οι εθνικές αρχές δεν είναι τόσο σίγουρο ότι μπορούν να τις ε, χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει να αποφύγουμε κινδύνους. και θα είχε σημασία για την ευρύτερη κατηγορία των ε, δικαιούχων. Αυτά ενέχονται στον κανονισμό για τις απλοποιημένες συνθήκες ε, οι επιλογές κόστους θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν καταποκοπήν ποσά και αν υπάρχουν να μην την χάνουν ελέγχου. Τέλος, ως προς τον καινοτόμο χαρακτήρα του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ δεν είναι καινοτόμο τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια μέσα στα πλαίσια του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Ε, εμείς το, με βλέπουμε σε αυτές τις πέντε χώρες δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα ότι άλλες χρησιμοποιούν το, L, το ΕΚΤ, Άλλε στο άλλο ταμείο. Δηλαδή βλέπω ότι όταν υπάρχει καινοτομία δεν ε, την χάνει χρηματοδότησης αποκλειστικά από το ΕΚΤ σε αυτές τις χώρες. Ως προς τη διατήρηση θέσεων εργασίας έχει σημασία, αλλά τη στιγμή που ο δείκτης ανεργίας έφτασε και το 40% σε μερικές, σε μερικές χώρες, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί για τους ε, Ρωμά βλέπουμε ότι φτάνουμε και μέχρι 50 και 60%. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και πολλές φορές δεν αρκούν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Αλλαγή Προεδρίας. Λοιπόν, στον Ερή Κετιέν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να δώσω τον λόγο για να απαντήσει μέσα σε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές είναι ερωτήσεις που ακούστηκαν και γραπτός υπέβαλα στην γραμματεία κάποιες απαντήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα σε στο χρόνο που έχω δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πολλές περισσότερες πληροφορίες λοιπόν στο σημείωμα το οποίο υπέβαλα. Πολλές ερωτήσεις όσον αφορά την πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο. Όντως σας είπα ότι στη Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στην Πουατού Σαγόντα έχουμε ένα 80% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ένα 20% μόνο τυχαίνει διαχείριση από την κεντρική διοίκηση. Και κατά αυτόν τον τρόπο συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εταίρους σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με όλους τους εξειδικευμένους ε, οργανισμούς, οργανισμούς διαμεσολαβητές θα έλεγα, όπως οι οργανισμοί για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την στέγαση κτλ. Όλοι ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα αυτά, επομένως οι τοπικές εταιρικές σχέσεις υπό την εποπτεία του νομάρχη της περιφέρειάς μας χρησιμοποιούνται, ενθαρρύνονται σε αυτό το περιβάλλον. Ναι λοιπόν, η πολιτική μας έχει αυτόν τον εδαφικό χαρακτήρα και προφανώς προωθεί όμως τα γενικά συμφέροντα βασική μας αρχή είναι να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που αποφέρουν αποτελέσματα. Μία ελερώτηση είχε να κάνει με τους κοινωνικούς δείκτες. Αναφέρθηκα εγώ σε κάποιους δείκτες αποτελεσμάτων. Όπως είπα όμως και η συγγήτρια θα ήταν ίσως καλύτερη, ενώ θα ήταν πιο θετικό να γίνει μια πιο συγκεκριμένη αποτίμηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία προσανατολισμού που να έχουν να κάνουν με όλον τον ε, πληθυσμό και να ουσιαστικά έχουμε προγράμματα τα οποία να βοηθούν τους ανθρώπους όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είτε πρόκειται για τους νέους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, είτε πρόκειται για πιο ηλικιωμένου πολίτες οι οποίοι θέλουν να υποφεληθούν κάποιων προγραμμάτων κατάρτισης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε τέτοια προγράμματα και να δούμε επίσης πόσοι συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Και επίση θα ήταν καλό να έχουμε και μια αξιολόγηση όσων έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα αυτά. Όσον αφορά τη μείωση των αναλφάβητων, νομίζω ότι έχουμε θέσει συγκεκριμένου στόχου και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία σα έδωσα πριν από λίγο θα ισχύουν είτε για την Πατού είτε για όλη τη Γαλλία και προφανώς περιμένουμε ότι θα έχουμε μία μείωση των, των αλφαβητισμού. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα για παράδειγμα στο σχολείο ή στις επιχειρήσεις, τον, την αγορά της εργασίας. Έχουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε σε κάποιες ε, τοπικές αποστολές από συγκεκριμένους εκπροσώπους. Δηλαδή να έχουμε κάποιους ε, εκπροσώπους οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες και να προτείνουν τα συμβόλαια αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ζήτημα τώρα της ε, απλούστευσης. Ζήτημα το οποίο προκύπτει φαντάζομαι πολύ συχνά. Δύο ιδέες θα ήθελα να φέρω εδώ πέρα. Δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό με τα δημόσια χρήματα. Στην παρουσίαση μου όμως είπα ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια μικρά προγράμματα. Και ο Γερμανός συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο, δηλαδή να έχουμε μία διάρθρωση διότι πολύ συχνά έχουμε διάρθρωση σε κάποια προγράμματα η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη απλούστευση σε κάποια προγράμματα, να έχουμε κάποια άλλα προγράμματα τα οποία θα έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Αναφέρομαι πάντα σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Να υπάρχει επίτε ένα εγχειρίδιο το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι φορείς υλοποίησης ε, των έργων, των προγραμμάτων ή οι αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων, είτε είναι εθνικές είτε είναι αποκεντρωμένες. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε περαιτέρω να εξετάσουμε τις ιδέες αυτές. Και τέλος, έρχομαι στο τελευταίο σας ερώτημα όσον αφορά το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το φαινόμενο μόχλευση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερους πόρους ξεκινώντας από την κοινωνική ενσωμάτωση, θα μπορούσαμε να έχουμε υψηλότερους σπόρους στο μέλλον ή να προβλεφθούν και κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις, την αιρεσιμότητα. θα μπορούσαμε μια κάποια διακύμανση στα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται να έχουμε και πιο θετικά συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου και να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τελικά τα καλά προγράμματα κατά αυτόν τον τρόπο. Απάντησα, φαντάζομαι, στι περισσότερε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο προσκεκλημένο, θα ήθελα να σας ε, θέσω μία ερώτηση σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί έγινε μία ανάλυση της λειτουργίας του ΕΚΤ και μιλήσαμε για δυσκολίες που υπάρχουν. Υπάρχουν ε, αντιδράσεις ως προς αυτό το θέμα. Θα ξαναλάβω το λόγο λοιπόν. Πράγματι στο Πουατού έχουμε 14 οργανισμούς μεσολαβητές για ενώ για τα λειτουργικά προγράμματα 17. Προσπαθούμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε. Το ελεγκτικό συνέδριο ζητά ε, να γίνει εξορθολογισμός έτσι ώστε να ε, υπάρχουν επιδοτήσεις από το ΕΚΤ. Θα πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Νομίζω ότι οι τρεις άξονες οι οποίοι προαναφέρεται ε, συζητούνται από το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κοινωνική συμμετοχή. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα χάσουμε μέσα σε μία πολυπλοκότητα οργανισμών και πολλών οργανισμών κυρίως. Θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν, υπάρχει και ο ΑΕΔ και οι ενδιάμεσοι οργανισμοί και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να, να αναγνωρίσουμε τις καλές πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικές και μετά να ορίσουμε μία, ένα πλαίσιο εργασίας έτσι ώστε να δούμε ε, κατά πόσο είναι επισφαλής οι εργασίες. Ευχαριστούμε. Μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις επικρίσεις του ελεγκτικού ε, συνεδρίου σε σχέση με το, τη λειτουργία αυτή. Ο κύριος Κούλμαν έχει το λόγο. Α, έχετε άλλη σειρά, εντάξει. Okay, vielen Dank. Ich äh, möchte gern zu drei Bereichen Ο κύριος Μπάρτελς ε, θα ήθελα να αφαιρθώ στην εταιρική σχέση, την, ε, τους κοινωνικούς δείκτες και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε εργαστήριο. Όσον αφορά την εταιρική σχέση, σίγουρα θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ίση μεταχείριση σε όλες τις περιοχές. Να η απάντηση που έχω να δώσω. Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, το βλέπουμε και στη Γερμανία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διασπάσουμε τις υφιστάμενες δομές. Θα πρέπει να γίνει αυτό με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ορισμένες ε, φορές υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν θέλουν να συνεργαστούν με επιπλέον φορείς. Θεωρούν ότι ε, η υφιστάμενη δομή είναι επαρκής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πού βρίσκονται οι ενδυνάμοι φορείς, οι ενδυνάμοι εταίροι που θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να δημιουργήσουν επιτόπου τη θέμενη αξία. Όσον αφορά τώρα τους κοινωνικούς δείκτες, Στη Γερμανία είδαμε τι προτείνει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και θέλαμε να δούμε αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλέον δεδομένα, δηλαδή να πούμε ποιο είναι το ποσοστό των μακρόχρονα άνεργων, οι οποίοι όντως είχαν μείνει για ένα πολύ χρονικό διάστημα εκτός εργασίας Έχουμε τις πληροφορίες αυτές από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αλλά αυτό από μόνο του δεν έφτανε ως κοινωνικός δείκτης. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι μακροχρόνια άνεργοι για τους ε, οποίους πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα προκειμένου να τους βοηθήσουμε και όχι απλώς να τους αξιολογούμε ή να τους δίνουμε κάποιες ε, καταποκοπήν λύσεις χωρίς όμως να υπάρχει μια καθοδήγηση για τους ανθρώπους αυτούς, χωρίς να υπάρχει μια πλαισίωση για αυτούς τους πολίτες. όσον αφορά αυτή την δεξαμενή απασχόλησης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Γερμανία οι οποίοι όντω εργάζονται, αλλά δεν καταφέρουν να ζήσουν από την εργασία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι για του ανθρώπου αυτού θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, αν πραγματικά θέλουμε να του επανεντάξουμε ουσιαστικά στην αγορά εργασία. Επί του παρόντος δεν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση προκειμένου να εφαρμοστούν τέτοιες αποφάσεις και όσον αφορά την ε, ανεργία, μα, συγγνώμη, την απασχόληση υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες, όπως για παράδειγμα ένας δείκτης ικανοποίησης, την ε, δυνατότητα δημιουργίας περαιτέρω θέσεων εργασίας. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι σε μια πρόσφατη έκθεση υπόθηκε ότι η Γερμανία υστερεί ότι έχει κάνει λίγα πράγματα τελικά στον τομέα τη απασχόληση Και όσον αφορά το ζήτημα τη απασχολησιμότητα, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κάποιε απομονωμένε λύσει χωρί να υπάρχει όμω μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική, κυρίω για τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Όσον αφορά τώρα την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ένα εργαστήριο πειραματισμού προκειμένου να προκύψουν κάποιες νέες ιδέες. Εργάζομαι πολλά χρόνια στη θέση την οποία κατέχω και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πλέον σε θέση να αναπτύξουμε και νέα προγράμματα. Δηλαδή να έχουμε τέτοιες δομές όπου θα έχουμε και νέους και πιο ηλικιωμένους, ότι θα υπάρχει μία μεταφορά γνώσεων από τη μία ηλικία στην άλλη, ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Δεν νομίζω επίση ότι μπορούμε αυθαίρετα να θέσουμε ένα έτος ταξιοδότηση, όπως για παράδειγμα το έτος των 67 ετών. Νομίζω, κυρίως αν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο όριο ταξιοδότηση πανευρωπαϊκά, θα καταλήξουμε σε περιπτώσει που πάρα πολλοί άνθρωποι θα εγκαταλείπουν τη δουλειά του απλώ νωρίτερα, προτού φτάσουν δηλαδή στην ηλικία αυτή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε του ανθρώπου στη θέση εργασία του, ακόμα και όταν οι άνθρωποι αυτοί γυράσκουν. Θα πρέπει όμως να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο η οθέτηση των μέτρων αυτών χωρίς να υπάρχει μια στρέβλωση της αγοράς εργασίας ή χωρίς να δημιουργηθούν επισφαλείς θέσεις εργασίας. Από γερμανικής πλευράς νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα συγκεκριμένο. Το μόνο που λέμε είναι να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, μένουμε στα λόγια, δεν προχωράμε στις πράξεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα αυτά. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να δώσω το λόγο και στην Επιτροπή. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει από πλευράς Επιτροπής Ονομάζομαι Αντριάννα Τόσεβα από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ασχολούμαι με τη μελλοντική νομοθέτηση, την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Σας ευχαριστώ γιατί μας καλέσατε σήμερα και ακούσαμε τη θέση ορισμένων από τους δικαιούχους, ε, εκείνων που χρησιμοποιούν πραγματικά το ΕΚΤ Έχω καταγράψει τα σαφή μηνύματα των τριών συναδέλφων, έτσι ώστε το ΕΚΤ να βρίσκεται στη θέση που του αρμόζει, γιατί στην παρούσα κατάσταση την οικονομική και κοινωνική θα πρέπει να κάνουμε πολλά για τους ε, ανθρώπους στην Ευρώπη. Όσοι είδατε τον γενικό κανονισμό, τις κοινέ ε, διατάξεις και τον κανονισμό του ΕΚΤ, Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή έχει πραγματικά δεσμευτεί να ε, ασχοληθεί για την ισότητα των δύο φύλων και την έλλειψη διακρίσεων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με δράσεις που σχετίζονται με τις επιμέρους δραστηριότητες του ΕΚ οι σχέσεις εταιρικότητας θα πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως θα πρέπει να δούμε τι πόρους έχουμε στη διάθεσή μας και πιστεύουμε ότι το ελάχιστο 25% δηλαδή το 25% είναι το ελάχιστο, θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλότερο, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη σχέση εταιρικότητας εκεί όπου μπορούμε και να έχουμε και έναν ε, κώδικα συμπεριφοράς έτσι ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει επί τόπου από το ΕΚΤ για να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πραγματικά δικαιούχοι. Ως προς τις πληρωμές αναφερθήκαμε στην ανάγκη σωστών ε, πληρωμών στον οργανισμό για τις κοινέ διατάξεις έχουμε προτείνει οι πληρωμές να εκτελούνται από, τις, από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη μόνο όταν έχουν γίνει από τη διαχειριστική αρχή στον τελικό δικαιούχο. Θέλουμε ε, οι αιτήσει πληρωμών να πιστοποιούνται εγκαίρως και να καταβάλλονται και να καταβάλλονται υποστηρίζουμε την ανάγκη να έχουμε καλούς, σαφείς δίκτες για να έχουμε εικόνα των επιπτώσεων του ΕΚΤ για τους νέους, για τους ηλικιωμένους, για τους φτωχούς και για τους αναξιοπαθούντες. Και δεν είχαμε επαρκείς δείκτες μέχρι τώρα για τις μελλοντικές δράσεις. Το ΕΕΛΚΤ θεωρείται και ένα κοινωνικό εργαστήριο όπου μπορούμε να προβάλλουμε νέες δράσεις για το μέλλον και μπορούν να το κάνουν και οι πολιτικοί αυτό και πιστεύουμε ότι ορισμένες από τις κοινωνικές καινοτομίε από το ΕΚΤ οδηγούν σε αλλαγές πολιτικών στα κράτη-μέλη. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο αφορά την έλλειψη διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες στη, στον κανονισμό κοινών διατάξεων για να αποτιμήσουμε τα λειτουργικά προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα, για να δούμε ποια είναι τα επιμέρους ποσά τα οποία μπορούν να κατανεμηθούν. Μου έκανε και εντύπωση το σχόλιο του ελεγκτικού συνεδρίου στη Γαλλία για τους ενδιάμεσους οργανισμούς. Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερο streamlining και όταν υπάρχουν ενδιάμεσοι οργανισμοί, οι οργανισμοί αυτοί να μην είναι ενδυνάμοι δικαιούχοι. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι οργανισμοί και ποιοι μπορούν να είναι οι δικαιούχοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ δικαιούχων και ενδιάμεσων οργανισμών. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ε, περιμένουμε και την γνωμοδότησή σας. Πρόεδρος να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή. Φτάνουμε στο τέλος των εργασιών μας, αλλά νομίζω ότι κάτι θέλει να μας πει ε, εν συντομία αυτά που θέλει, γιατί πρέπει να φύγουν οι διερμήνες. Θα ήθελα εξ ονόματος ε, των συναδέλφων, σκιωδών και ε, μελών να πω ότι υπάρχουν μεγάλα κίνητρα για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ και τους πάνελιστ. Πρόκειται για την τελευταία μας ακρόαση για το ΕΚΤ. Είναι ένα θέμα που ήδη μας είχε απασχολήσει ως προς την ανάγκη κοινωνικού διαλόγου για να προωθήσουμε τις δραστηριότητες του ΕΚΤ και να δώσουμε ένα κίνητρο στα σχέδια αυτά. Η κοινωνική εταιρικότητα μας βοηθά για να ορίσουμε αυτούς τους πολιτικούς στόχους μέσω σχεδίων. Θα πρέπει όλοι να συμπεριλαμβάνονται και να είναι κοινωνοί όλων των σχεδίων για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να προωθήσουμε και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο ε, ενεφανίστη αφορά τις πολιτικές, την, πολιτική, ε, την ευρωπαϊκή πολιτική που θα πρέπει να συντονιστεί με τις εθνικές ε, πολιτικές. Εάν υπάρξει ρήξη σε αυτή την αλυσίδα δεν θα τα καταφέρουμε. Επίσης υπάρχει ανάγκη απλούστευσης. Μίλησα για την έννοια του κατοφλίου της διαφοροποίησης των θεμάτων, την αποτελεσματικότητα των ενδιάμεσων οργανισμών και εδώ βλέπουμε ότι στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάρχει, υπάρχουν περιθώρια προόδου, μεγάλης προόδου. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά που μας επιτρέπει το ΕΚΤ μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής καινοτομίας και όπως όλοι είπατε, ένα από τα προβλήματα της αποτελεσματικότητας του ΕΚΤ αφορά τους φτωχότερους και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εξατομικεύσουμε τις ανάγκες, διότι πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε καλά μέσα στα πλαίσια αυτής της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε θάρρος και εμείς και η κοινωνικοί εταίροι. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους. Ε, λυπάμαι που δεν σας άκουσα όλους γιατί έπρεπε να λείψω από την αίθουσα. Το επόμενο, η επόμενη φάση είναι η έκθεση Μωρέ στις 22, 23 ή 23-24 Απριλίου. Τελειώσαμε τις εργασίες μας σήμερα και θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί για τη συνέχεια των εργασιών μας. Χαίρετε.